Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καθίστε σας παρακαλώ, διότι έχουμε μια μικρή καθυστέρηση που δεν πειράζει, αλλά μην γίνει μεγάλη. Ε, δεχτείτε τη συγγνώμη του κυρίου Τόιρερ που κολλείται και απουσιάζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ εγώ για να το αναπληρώσω. Πρώτο θέμα. Έχετε σχόλια για τη μέση διάταξη, συμφωνείτε να την εγκρίνουμε. Άρα εγκρίνεται. German Παρακαλώ τους Γερμανούς φίλους πριν κάνουν το μεγάλο συνασπισμό να προσέξουν λίγο να συνεδριάσει η Επιτροπή μας. <laughs> Okay, let us start from voting. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Έχουμε την κυρία Ινέσα Γιάλα Σέντερ παρούσα. Γιατί είναι δική της η έκθεση. Next report would be... Καλά, επόμενη έκθεση τότε. Α, και αυτή τη συνέση είναι. Ε, τότε να φτάσουμε στον κύριο Πίπερ. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά. Opinion, and then Mr. Geyer's opinion, and then we can... We can... Λοιπόν, παρευρίσκεται ο κύριος Γιένς Γκάιερ και έχουμε και δική του γνωμοδότηση να ψηφίσουμε. Συμφωνείτε να αρχίσουμε από αυτή. Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν. Παράγραφος πρώτη, τροπολογία πρώτη της κυρίας Γκρέσλε. Ψηφίπε in Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. item, 6. We are voting the list of uh, Mr. Geyer's opinion. Draftsman Jens Geyer. Λοιπόν, είπαμε ότι συντάκτης νομοδότησης είναι ο κύριος Jens Geier έλεγα να δείξουμε μια ευελιξία. Οι παρόντες ε, συντάκτες ε, να βλέπουν την έκθεσή τους να ψηφίζεται. Ήρθε η κυρία Ινέσα Γιάλα, αλλά έχουμε αρχίσει με την άλλη έκθεση. Ε, παράγραφος 5, τροπολογία 2, Γιάν Μέλντερ, ψηφί Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Μέλντερ. Η τροπολογία 3 του Μπαρτ Στάς, ψηφί κατά ένας αποχή εγκρίνεται σας ευχαριστώ η τροπολογία 4 του κυρίου Πίπερ ψηφίπε. κατά αποχές εγκρίνεται 5 πάλι του κυρίου Πίπερ ψήφι κατά άποχες έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση ε, Voting, vote is closed. Πέρας τις Εγκρίνεται. Τροπολόγια παριθμών 6 και 7 της κυρίας Γκέσλε, Γκέσλη. Κατά. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία όπως και προηγουμένως. Η τροπολογία παριθμών 8. Ψηφί υπέρ. Την 7 την ψηφίσαμε. 8 λέμε. Ψήφι υπέρ. κατά άποχες εγκρίνεται. Vote on the draft opinion. Το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε, το σχέδιο γνωμοδότησης μάλλον, κατά, όχι, ηλεκτρονική διορθώνει ο πρόεδρος, αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. Αφού έφτασε και η Ινές Αγιάλα, μπορούμε να ψηφίσουμε τη δική της νομοδότηση. Με ποια σειρά, γιατί έχει δύο. Το GNSS πρώτα. Λοιπόν, στην αιτιολογική σκέψη 8 έχουμε την τροπολογία παριθμών 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογική υπερθών 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. open. Άρχεται η ψηφοφορία. Και τελειώνω. Απορρίπτεται. 12 του Ζων Πιεροντή ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 Υπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τσεκ. Καλά. Ας την ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία είναι. 15, συγγνώμη, είπε. Κατά. Όχι, 14 διορθώνει ο πρόεδρος. Ε, ε κατά. Αποχές έλεγχος. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 14 ήταν αυτή, έτσι, ωραία. 15 τώρα. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί. Όχι. ψηφίτε. Κατά. Απόχες. Απορρίφτεται. Με μικρή διαφορά. Θέλετε ξανά έλεγχο. Ξανά λοιπόν. Τη 15 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 15, 16 και 17 μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Vote is closed. Ε, πέρας. Απορρίπτονται. Βλέπετε, καμιά φορά έχει δίκιο και ένας άπειρο σχετικά πρόεδρος. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατά την ταπεινή μου άποψη. Θέλετε να το ελέγξουμε, όχι. Η 19 ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. 20 υπέρ Τσεκ. Για τη 19. Ας την ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. πολύ μικρή διαφορά. Παρ' όλα αυτά απορρίπτεται. 20. Ψήφι Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Η τροπολογία 21 ψηφίπε. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Λυπάμαι, αλλά περίφθη. Τροπολογία 2 ψηφίπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Ψήφι υπέρ. Είναι συμβατή με την προηγούμενη. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαρινέσκου. Η 3. Ah, Α, ah, όχι, καταπίπτει σε περίπτωση που εγκριθεί 24, λέει εδώ. Ναι. Η 4 είπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 25 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική παρήθευση καλώς. Για την 25 αρχίζει τώρα. Λήξεις. Απορρίπτεται. Ποια ήταν αυτή η 25. Ερχόμαστε στην 5 τώρα λοιπόν. Τροπολογία έρθουμε, 5 ψήφι πέρα. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 26. 7 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία είναι πέρα. κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 27 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 28 είπε, κατά άποχες εγκρίνεται 29 είπε, κατά άποχες εγκρίνεται λοιπόν τελική δεν έχουμε α έχει εδώ μια προφορική της εισηγήτριας στην τροπολογία 18 εγκρίθηκε Α, εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Τελική ψηφοφορία Will Be, uh, let us make electronic vote. Ηλεκτρονικά πρέπει να γίνει αυτή. Αρχίζει τώρα. Πέρασε. Okay, what is still coming? Congratulations. Συγχαρητήρια. Κανείς δεν καταψήφισε η μία αποχή. Συγχαρητήρια στη συντάκτρια της νομοδότησης. Πάλι της κυρίας Ινές Αγιάλα Σέντερ πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Λοιπόν, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Τροπολογία. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 21. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 23. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κατά τη γνώμη μου αλλά σε παληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία Τέλος. Απορρίφθηκε όντως. 27, τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. 29 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε καλύτερα Αρχίζει η ψηφοφορία. Πρόκειται την τροπολογία 31. Τέλος. Απορρίφθηκε. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτή 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 68 υπέρ Α, και οι 74 μαζί 68 και 74 μαζί υπέρ κατά αποχές κατά τη γνώμη μου απορρίπτονται θέλετε επαλήθευση ναι. Καλά λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίφθηκε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές. Ίσως με μια ψηφοδιαφορά προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Ας επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίφθηκε ωστόσο. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ίσως επαληθεύσουμε. Ωραία. 36 αρχίζει η ψηφοφορία. Είστε υπέρ ή κατά. Πέρας. Απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα ας αρχίσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Παρακαλώ λοιπόν στο μέλλον να σηκώνετε καλά τα χέρια. 39. Υπέρ. Κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά αλλά ας ε, επαληθεύσω τέλος Α, με δύο ψήφους διαφορά. Απορρίπτεται λοιπόν η 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 41 απερίφθη ρωτάει κάποιος μάλιστα 41 λοιπόν όλες μαζί μέχρι και την 46 μέχρι την 46 ψήφι υπέρ κατά αποχές Θα κάνουμε επαλήθευση ωστόσο. <laughs> Πέρας. Απερίφθησαν αυτές. Προφορική τροπολογία Α της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, υπέρ. Νέο άρθρο 27. Βλέπω ότι γνωρίζετε το αυτό. Υπέρ λοιπόν κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Κατά. Ε, συγγνώμη, υπέρ, υπέρ, με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται και μάλιστα σαφώ. Τροπολογία 70 μέχρι τι 73 όλες μαζί, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Σας ευχαριστώ, έτσι προχωρούμε και πιο γρήγορα κάπως. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ 75 μέχρι... μέχρι... Α, οι δύο αυτές, 75-76. Καλά λοιπόν. Μαζί αυτές οι δύο, 75-76, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται και σας ευχαριστώ. 53 έως 56. Νομίζω μπορούμε να τις πάρουμε αυτές όλες μαζί. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 77 αυτή πρέπει να ξεχωριστά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 και μάλλον μέχρι την τροπολογία 5, αν συμφωνείτε όλες μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 6 και 7, 8. Όλες μαζί γίνεται. Όχι, χωριστά, καλά λοιπόν. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Ο κύριος Μπράντμπουρν έπρεπε ένσταση για την ψηφοφορία όλων μαζί. 7 7 υπέρ μόνο για την 6 ε, προέβαλα ένσταση για να συζητηθεί, να ψηφιστεί με τις άλλες. Άρα τότε λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, ε, α, α, τώρα προβάλλει ένσταση η, η 7 και 8 λοιπόν μαζί γίνεται, ναι. 7 και 8 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε καλύτερα 7 και 8 τέλος μία ακόμη ε, ψήφος κατά. Καλά, έχει απορριφθεί λοιπόν, εντάξει. Τροπολογία 9, 10 κλπ. έως 14. Αν συμφωνείτε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Αιτιολογική σκέψη 17 με ψήφο κατά τμήματα. Πρώτο μέρος, προσθήκη, έγκριση μέτρων κλπ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 23 με προφορική τροπολογία της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 16 εκπίπτει. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση. Μετά 17, 18, 19, 20 και 2. Όλες μαζί. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη που είστε τόσο ευγενείς ε, και δεχτήκατε υπέρ κατά αποχές ψηφίστηκαν και απορρίφθηκαν ομού. Τώρα η τελική ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφος μία δική σας υπέρ κατά. Μάλιστα, ωραία. 16 λοιπόν υπέρ και μία ψήφος κατά συγχαρητήρια. Τώρα προχωρώ στην έκθεση του αξιότιμου κυρίου Ριβελίνη και πρώτη τροπολογία υπάρχουν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 εδώ προβλέπεται ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά ας επαληθεύσουμε αυτός τέλος δεύτερο τμήμα της 6 Είστε λοιπόν εσείς υπέρ κύριε Κλίντς. Ωραία. Αυτά λοιπόν εγκρίθηκε. Λοιπόν, 7 υπέρ κατά. Αποχές. Ας, ας υπαλληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. 8, 8 και 1. Μια σημεία δηλαδή. Ε, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζετε ότι απαιτείται επαλήθευση Ας αρχίσει η ψηφοφορία. Νομίζω η κυρία Γκρέσλε δεν σηκώσει το χέρι της. Απερίφθη λοιπόν τώρα που έληξε η ηλεκτρονική ψηφοφορία και είδαμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Τροπολογία 10. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται σαφώς. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται και αυτό το τμήμα. Α, κάποιος ζητεί επαλήθευση. Καλώς λοιπόν, ας αρχίσει η ψηφοφορία. Τέλος. Εσάς κύριε Κλίντς είστε υπέρ. Καλά, ευχαριστώ λοιπόν που στηρίζετε. Ε, το τρίτο τμήμα τώρα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται και αυτή. Α, ίσως όχι. Α, εγκρίνεται, έχετε δίκιο. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 λέει ο πρόεδρος. Α, όχι, 4 είναι το σωστό. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται αυτή. Τελική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Συγχαρητήρια. 16 υπέρ και δύο μηδενικά για τα υπόλοιπα. 17-0-0 λέει ο πρόεδρος. Πολύ καλό αποτέλεσμα κύριε Ριβελίνη Συγχαρητήρια. Και επανέρχομαι. Επανέρχομαι λοιπόν στην άλλη έκθεση της κυρίας Σεντέρ. Λοιπόν, ψηφοφορία άρχεται για την τροποποίηση του κανονισμού GNSS. Ψηφίσατε, τελείωσε. Σας ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα λοιπόν μαζί μας ε, τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη απουσία του κυρίου Καλτέρα ίσως. Είχε προσγειωθεί όταν ξεκινήσαμε, είναι θέμα λεπτών. will not arrive Φτάσατε στην ώρα σας, Πρόεδρε και Καλδέρα. Perfectly on time. So, item, welcome, President Caldera. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Πρόεδρο Καλδέρα. Αναφέρομαι στο 8ο θέμα, μελλοντικό ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου, η συγγήτρια είναι σαν Αγιάλα Σεντέρ. Ινές, θέλεις να ξεκινήσεις. Ναι, θέλω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτή την έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Δυστυχώς μόνο στα αγγλικά υπάρχει προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει σε λίγες γλώσσες. Τι θέλω εγώ με αυτή την έκθεση να κάνω. Να αρχίσει η συζήτηση στην Επιτροπή μας προς τη βελτίωση των ε, μέσων ε, που έχει στη διάθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα για να ελέγχει, να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να προτείνει τα απαραίτητα μέτρα τελικά έτσι ώστε να βεβαιώνονται πάντα οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι είναι χρηστή η χρήση των κοινοτικών πόρων, των χρημάτων των φορολογουμένων, δηλαδή να γίνεται σωστή εκτέλεση, να πιάνουν τόπο τα χρήματα, να επιτυχάνονται οι στόχοι και πάντα στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων ή των μελημάτων αλλά και των ανισχυών των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό με ενδιαφέρει, βελτίωση λοιπόν των μέσων και εδώ το ελεγκτικό συνέδριο ανέκαθεν ε, ήταν μεγάλη υποστήριξη και θαυμάσιο συνομιλητή μα. Πολλές φορές οι συζητήσει ήταν συναρπαστικές και με μεγάλο πάθος, γιατί πάντα ε, του ενδιαφέρει να γίνεται καλή χρήση των κοινοτικών πόρων και πάντα ε, σε νόμιμα πλαίσια, σε θεμητά και να πιάνουν τόπο, είπαμε, και να είναι αποτελεσματικά. Αλλά ταυτόχρονα συνεργαστήκαμε με το ελεγκτικό συνέδριο για να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει Που είδαμε ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μα έχει φέρει νέα δεδομένα και προκλήσει που πηγαίνουν ακόμα ε, πιο πέρα από τα ιστορικά ε, μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας. Είχαμε λοιπόν μια σειρά από με το ελεγκτικό συνέδριο και εδώ στην Επιτροπή μας και αλλού και στην Επιτροπή λοιπόν Ελέγχου του Προϋπολογισμού είπαμε ότι θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία στην έκθεση αυτή όπως θα δείτε. Το πρώτο είναι ο γενικός ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου, πώς έχουμε συνεργαστεί και πώς μετά από τόσες πολλές συζητήσεις μπορούμε να φανταστούμε το μελλοντικό ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Να υπάρξει μια αλλαγή περισσότερο ή λιγότερο βαθιά, δεν ξέρω. Ε, ξέρω ότι σιγά σιγά το ελεγκτικό συνέδριο έχει αλλάξει ήδη και το ένα δεύτερο στοιχείο είναι ο διορισμός των υποψηφίων ε, μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί στο παρελθόν είχαμε προβλήματα, περισσότερο λιγότερο σοβαρά. Βρέθηκαν κάποιες λύσεις, αλλά τελευταία και στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικά ως θεσμικό όργανο, έχουμε ανησυχήσει κάπως. Για να μην πω ότι έχουμε ενοχληθεί και θυμώσει με το Συμβούλιο. Παρά την αντίθετη ε, ε, δική μας άποψη ε, για το διορισμό ενός υποψηφίου, το Συμβούλιο μας παραγκόνησε και τον διόρισε. Έτσι κι αλλιώς. Yo creo que lo que propuesto se ε, πάντως μπορούν να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες και το πρώτο μέρος της έκθεσής μου τι προσπάθησα να κάνω. Είχαμε πολλές συζητήσεις και φτάνουμε περίπου στο τέλος της θητείας προσπάθησα να θέσω νέες προτεραιότητες. Αναγνωρίζω βέβαια τη σημερινή ε, δουλειά του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά θέλω να του δώσω περισσότερη έμφαση, περισσότερη ορατότητα. Ναι. Δηλαδή, από την αρχή του προγραμματισμού, δηλαδή των εργασιών των διαφόρων θεσμικών οργάνων, θα πρέπει να συμμετέχει το ελεκτικό συνέδριο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το ετήσιο πρόγραμμα και για το πολιετές πρόγραμμα. Γιατί χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία, την πείρα, τις ικανότητες εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων που μπορεί να κάνει το ελεκτικό συνέδριο. Για ποιο τεχνικά ζητήματα μιλώ τώρα ως προς τον έλεγχο και πώς μπορεί από την αρχή να βελτιωθεί. Γι' αυτό λοιπόν η προτεραιότητα για μένα είναι ως εξής. Υπάρχει ανάγκη το ελεγκτικό συνέδριο από την αρχή να συμμετέχει από τη φάση του προγραμματισμού με ε, επιμέρους και επίκαιρες νομοδοτήσεις από την αρχή να συνοδεύει αυτή την προσπάθεια. Ήδη έχει γίνει ε, μια τέτοια προσπάθεια και το αναγνωρίζω και ο πρόεδρος Καλντέρα εδώ πραγματικά ε, βοήθησε πολύ. Ε, κάθε φορά λοιπόν που και λόγω της κρίσης προσπαθούσαμε να ξαναβρούμε και κάποια άλλα μέσα και τρόπους χρηματοδότησης και θέλησε και το ελεκτικό συνέδριο να ξεπεράσει λίγο το ρόλο, το κλασικό του εκ των υστέρων ελεγκτού τα λοιπά και εκ των προτέρων να μπορεί να γνωμοδοτεί, να μας λέει τη γνώμη του έτσι ώστε αυτά τα νέα μέσα να συνοδεύονται και ε, από τα απαραίτητα ελεγκτικά εργαλεία. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ ουσιαστική ακόμα αυτή η προσπάθεια. Σε μεγάλο βαθμό το ελεγκτικό συνέδριο έχει περιοριστεί σε ένα ρόλο ε, κλασικό, ελεγκτικό των επιδόσεων του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ένα δεύτερο που λέω στην έκθεσή μου είναι ότι τώρα έχουμε ανάγκη να εμβαθύνουμε όχι μόνο ε, το νομικό σκέλος ας πούμε και το νομότυπο πώς εκτελείται ο προεπολογισμός εντάξει ε, εκτελείται σε ε, σωστά πλαίσια και ανταποκρίνεται στο ρόλο του Αλλά θα πρέπει και ένα άλλο στοιχείο να αναλάβει το ελεκτικό συνέδριο, πέρα από τον κλασικό έλεγχο του προϋπολογισμού. Είναι πιο περίπλοκες αυτές οι εκθέσεις ως προς τις επιδόσεις και την απόδοση του προϋπολογισμού. Χωράει μεγαλύτερη συζήτηση εκεί, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες έτσι ώστε ο, ο κόσμος, οι πολίτες να καταλαβαίνουν όχι μόνο ότι σωστά και ορθά δαπανώνει τα χρήματα, αλλά ακριβώς για τους σκοπούς που έχουν αποφασίσει οι νομοθέτες. Δηλαδή, θα μας τα ε, πει και μας τα έχει πει το ελεκτικό συνέδριο ε, ότι ε, δεν υπήρχαν παρατυπίες, δεν υπήρχαν σφάλματα, δεν υπήρχαν απάτες μεν στην εκτέλεση κάποιου προϋπολογισμού, αλλά δεν επετέχθη ο στόχος, γιατί μπορεί να ήταν υπερβολικά φιλόδοξο ή μπορεί να ήταν κακά σχεδιασμένο το πρόγραμμα κτλ. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ελέγχουμε μόνο την νόμιμη και τη χρηστή διαχείριση, αλλά και την απόδοση τελικά ε, και τις επιδόσεις. Και τέλος, η δήλωση αξιοπιστίας που δεν θα μπορούσε άλλωστε να λείπει. Το ξέρω ότι είναι αυτό κάτι το οποίο οφείλει να παρέχει το ελεκτικό συνέδριο. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας έχουμε βρει όλες τις βέλτιστες πρακτικές, όλες τις συμβούλες, όλες τις οδηγίες. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η δήλωση αξιοπιστίας μπορεί να είναι ένα εργαλείο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό ή ο μοναδικός άξονας ή ο μοναδικός γνώμονας ο οποίο θα μετράμε τη δραστηριότητα του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα εργαλείο για μένα είναι παραπάνω. Μπορεί να ε, βελτιωθεί και να εξυγχρονιστεί. Δεν αντιλέγω και περιμένω να ακούσω και τους συναδέλφους προς την κατεύθυνση αυτή. Θα μπορούσαμε να το φανταστούμε και διαφορετικά, όχι μια ε, ετήσια ας πούμε τέτοια άσκηση ε, που απορροφάει τόση ενέργεια και τόσο κόπο από το ελεγκτικό συνέδριο ε, θα μπορούσε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, έτσι κάπως πιο κυκλικό ή βλέποντας και εντοπίζοντας πραγματικά που υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και που χρειάζεται να εμβαθύνει περισσότερο ο έλεγχος. Νομίζω με τα δύο προηγούμενα που προτείνω βελτιώνεται η λειτουργία του ελεκτικού συνεδρίου και θα πρέπει να ενημερώνεται και το ελεκτικό συνέδριο και να προσαρμόζεται με την πραγματικότητα της ζήτησης ε, από πλευρά ελέγχου. Για να καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος και άλλωστε αυτό αναμένει από εμάς. Λοιπόν, αυτά προτείνω στην έκθεσή μου. Δεν είναι δικές μου σκέψεις, δικές μου εφευρέσεις. Προσπάθησα να παρακολουθήσω και την εξέλιξη και την τάση που εμφανίζει το ελεκτικό συνέδριο και μετά από δική μας άλλωστε επιθυμία και αίτημα. Και προσπαθώ να του δώσω λίγο περισσότερη σάρκα και τα... κάνω μια προσπάθεια να αναδιατυπώσω τις προτεραιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου και να επιβεβαιώσω ε, τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει στο ελεγκτικό συνέδριο. Σεβόμενοι πάντα την ανεξαρτησία του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μας συνοδεύει από την αρχή, από τη φάση του προγραμματισμού το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν θα κάνει και το δικό του προγραμματισμό ως ε, ε, ανεξάρτητο όργανο. Και εμεί στο Κοινοβούλιο κάνουμε τη δουλειά μα, η Επιτροπή Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε θεσμικό όργανο έχει τον εσωτερικό του προγραμματισμό, αλλά όλα αυτά γίνονται πάντα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκών ε, προτεραιοτήτων που συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Φαντάζομαι και με τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε και τις καλές ιδέες που θα προκύψουν από το διάλογο θα καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε η ανεξαρτησία και η αυτονομία του ελεγκτικού συνεδρίου σε καμία περίπτωση να μην περιορίζεται από το γεγονός ότι ζητούμε ή απαιτούμε κιόλας να ε, εργάζονται από την αρχή και να συνεργάζονται μαζί μας στον προγραμματισμό. Έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα πρόβλημα που συνεχώς βρίσκουμε ε, μπροστά μας. Γίνεται ένας διάλογος κοφών. Εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε ένα είδος παρατηρητού ας πούμε και προσπαθούμε να μεσολαβήσουμε, να βελτιώσουμε τη συζήτηση και το διάλογο μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα αν δεν ξέρουμε από την αρχή ποια είναι τα απαραίτητα ε, μέτρα για τον έλεγχο αυτό, κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, ξέρω εγώ, που είναι απαραίτητη για να γίνει επιδόσεων αποδόσεων ή προγραμματισμού, τότε προφανώς ο διάλογος θα συνεχιστεί όπως έχει σήμερα. Συνεχίζει το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο και μετά μπαίνουν σε ένα διάλογο κοφών, κομισιών και ελεκτικό συνέδριο και έχουμε απογοήτευση και ματέωση. Αντί να υπάρχει συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δικαιολογήσει γιατί δουλεύει έτσι, γιατί έπραξε ως έπραξε, ε, ως θεσμικό όργανο στη δράση. Πάντα υπάρχουν μηχανισμοί έτσι, αμυντικοί. Και ε, αντίστοιχα και το ελεκτικό συνέδριο. Βάζει θέματα προθεσμίων, ε, διάφορα. Και έρχεται στη μέση το κοινοβούλιο που θα πρέπει να δώσει ένα πιο πολιτικό μήνυμα προς τους πολίτες και τελικά αισθάνεται κάποια απογοήτευση. Γι' αυτό λέω ότι το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει από την αρχή να συμμετέχει. Με την ανεξαρτησία του, με τις δυνατότητες που έχει, με την τεχνογνωσία του για να βοηθάει έτσι ώστε να αποφύγουμε και να προλαμβάνουμε πολλά προβλήματα. που μας τρώνε τόσο κόπο, τόση ενέργεια, τόσες συζητήσεις και στήρες μάλιστα, με πολύ μικρή πρόοδο. Πιο ενδιαφέρον δεν θα ήταν να μπορούμε από την αρχή να υπολογίζουμε στη συνεργασία του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τελικά αυτές οι γνωμοδοτήσεις του ελεκτικού συνεδρίου δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα έρχεται μόνο στην Επιτροπή μας Ελέγχου Προϋπολογισμού, που είμαστε έτσι κι αλλιώς ο φυσικός αποδέκτης και συνομιλητής, αλλά θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε και τις συζητήσεις σε άλλες επιτροπές, όπου ακριβώς συζητούν το προγραμματισμό και τους στόχους και καμιά φορά Είναι ενδιαφέρον ε, να το ξέρουν ε, οι επιτροπές. Για να μην απογοητεύεται και το ε, ελεγκτικό συνέδριο, γιατί ξέρω ότι πολύ συχνά κάνουν πολύ ωραίες μελέτες, νομοδοτήσεις κτλ που ε, άδοξα καταλήγουν στο κοινοβούλιο και περνούν απαρατήρητε, γιατί έχει άλλε προτεραιότητε στο κοινοβούλιο, άλλε δουλειέ κτλ. Έχει διαφορά φάσεω. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε, να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο για να καταλαβαίνουν καλύτερα οι πολίτε με ποιο τρόπο προσπαθούμε να εγγυόμεθα τη σωστή και καλή διαχείριση και εκτέλεση του προπολογισμού, να πιάνουν τόπο τα λεφτά και να ανταποκρίνονται και στι προτεραιότητε των πολιτών. Στο δεύτερο τμήμα όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται αρκετά περίπλοκες βασικά πρέπει να αναζητήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για συζητήσεις τις οποίες έχουμε ήδη κάνει είναι το θέμα του ορισμού των μελών. Είναι σαφές ότι για ένα νέο στάδιο, για μια νέα φάση εφόσον θέλουμε να υπάρξει ένα πιο αποτελεσματικό ανανεωμένο ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να σκεφτούμε μια κάποια νέα δομή. Θα πρέπει να δούμε και τι επιτρέπει η συνθήκη, τι μας λέει η συνθήκη. Το ελεγκτικό συνέδριο προβλέπεται να αποτελείται από ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος. Θα πρέπει να δούμε αυτή η πρόταση ακριβώς έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ολομέλεια αν θέλετε και ένα εκτελεστικό κομμάτι και ε, η Ολομέλεια θα αποτελείται από τους προέδρους των σωμάτων των ελεγκτικών συνεδρίων κάθε κράτους, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη θα ορίζει την εντολή του εκπροσώπου του κάθε κράτους μέλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει όχι μόνο τη μορφή συνεργασίας η οποία υπάρχει ήδη ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με τα εθνικά, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο, να εμπλέξουμε περισσότερο τα εθνικά ελεγκτικά ε, για τα θέματα της κοινή διαχείρισης και μέσα και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα προς τα οποία πρέπει να πιέσουμε ε, τις κυβερνήσεις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακριβώς ε, σε επίπεδο ελέγχου, επιδόσεων και τα λοιπά το κομμάτι της σύγχρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Αυτά για, το, για την Ολομέλεια το εκτελεστικό κομμάτι μειωμένο 9 ίσως μέλη, ο μέγιστος αριθμός. Εν πάση περιπτώσει εδώ θα ακούσουμε και, άλλοι, και άλλες ιδέες, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για 5 λοιπά Εγώ σκέφτηκα ένα μέγιστο αριθμό 9 εν πάση περιπτώσει έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπημένη εκπροσώπηση και των μεγάλων χωρών και των μικρών χωρών χωρίς να δημιουργηθεί κανενός ε, τύπου ε, επιφυλακτικότητα. Να υπάρχει λοιπόν μια ισορροπημένη σύνθεση και σε επίπεδο φύλου, κάτι το οποίο δυστυχώς ελείπει ιδιαίτερα σήμερα, και να προσπαθήσουμε αυτή την ανάμιξη που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στους επαγγελματίες ελεγκτές, στα μέλη τα οποία προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, από την έρευνα και τέλος θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον πολιτικό χώρο, χωρίς να ορίσουμε συγκεκριμένα όργανα, αλλά παρόλα αυτά να πετύχουμε ένα μείγμα θα έλεγα, το οποίο ε, δημιουργεί ακριβώς αυτό το σύνολο το οποίο λειτουργεί και σήμερα γιατί τη διαδικασία του ορισμού λοιπόν κάθε κράτος μέλος θα πρέπει ε, και αναφέρομαι στο εκτελεστικό κομμάτι τους ε, ανθρώπους τους οποίους προτείνει. Θα πρέπει επίσης το Συμβούλιο να κάνει και αυτό μία πρόταση, θα πρέπει ο καθένας να συζητά τις επιλογές αυτές επί τη βάση των κριτηρίων τα οποία έχει θέσει και να καταλήγουμε στις συγκεκριμένες προτάσεις, να δημιουργείται ένα short list τουλάχιστον δύο ανθρώπων, άνδρας γυναίκα, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μην κάνει ακροάσεις μόνο για ένα πρόσωπο, αλλά να υπάρχει δυνατότητα επιλογής και να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε λεπτομερώς το προφίλ ε, των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου και να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να απαλλαγεί το Συμβούλιο από την πιθανή αρνητική άποψη του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε πρόσφατα κάποιες αρνητικές εμπειρίες οι οποίες δεν θα πρέπει να επαναληφθούν. Παράλληλα νομίζω ότι η εικόνα των υποψηφίων σχετικά με αυτό θα πρέπει να έχει κάποια σχέση και με τα ευρωπαϊκά όργανα. Μπορεί να μας στέλνουν εξαιρετικούς εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Τράπεζα ή από το νιταφ αλλά πραγματικά δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή ανωση και πώς λειτουργεί πραγματικά. Είμαστε ένα ιδιαίτερο αν θέλετε σχήμα, λειτουργεί όμως με αρκετά θετικό τρόπο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να βελτιώσουμε τις μελλοντικές εργασίες του συνεδρίου. Λοιπόν, έκανα μια παρουσίαση των συγκεκριμένων σημείων όπως είπε το κείμενο είναι σχετικά περιορισμένο, ελπίζω μέσω των τροπολογιών να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε στο μέτρο του δυνατού και είμαι διαθέσιμη και ανοιχτή στα σχόλιά σας και στις προτάσεις σας. Thank you very much, Ευχαριστώ κυρία Σεντέρ. Εξαντλητική η παρουσίασή σας. Μία από τις προτάσεις σας έχει ήδη γίνει δεκτή το θέμα της ισορροπίας ανδρών και γυναικών και σήμερα η αντιπροσωπεία του συνεδρίου αποτελείται από μία γυναίκα και έναν άνδρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Καλντέιρα. Ε, σας ευχαριστώ που μας δίνετε την δυνατότητα να συνεισφέρουμε στην παρούσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ επίσης που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί θα πρέπει να φύγω σε αποστολή για ένα άλλο κράτος μέλος. Να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Γιάλα Σέντερ για την πρωτοβουλία της να προωθήσει τη συγκεκριμένη έκθεση. Η πρόταση κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του συνεδρίου, στη διοίκηση, στη διαχείριση και στο ρόλο του. Όπως γνωρίζω, εκτιμούμε την δυνατότητα την οποία μας δώσατε έτσι ώστε να μελετήσουμε τις προτάσεις σας θα σας ε, παρέχουμε, εφόσον επιθυμούτε, την άποψή σας για την πρόταση εκθέσεως ε, τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω ότι στην επόμενη συνάντησή σας της Επιτροπής σας με τα μέλη του Συνεδρίου, η οποία προβλέπεται στις 14, για τις 14 Οκτωβρίου, ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία Πάντως και σήμερα θα μπορούσα να σας δώσω τις αρχικές αντιδράσεις μου σε κάποιο από τα σημεία της έκθεσης ε, τα οποία βασίζονται ε, και στις παρατηρήσεις που έγιναν με τώρα σε ό,τι... Για το μελλοντικό ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου θέλω να πω το εξής. Ε, είχαμε πολλές ανταλλαγέ και μάλιστα η τελευταία ήταν την περασμένη εβδομάδα ακριβώ εδώ στην Επιτροπή σας. Κατά την άποψή μου ο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου θα πρέπει να ιδωθεί ε, στα πλαίσια των εργασιών ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου και στα πλαίσια της συνθήκης, γιατί λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διακυβέρνησή της κάποιες αλλαγές. Εμείς είμαστε ελεγκτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποιο είναι ο εποπτικός ρόλος του Κοινοβουλίου για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έτσι ορίζονται όλα αυτά από τη συνθήκη και δικός μας ε, ρόλος είναι να είμαστε εξωτερικός ελεγκτής. Αυτό τι σημαίνει. Θα πρέπει να δίνουμε ε, ε, προτάσεις για μια πολιτική ε, μορφή ελέγχου ενός θεσμικού οργάνου. Τα είπε η κυρία Γιάλα ακριβώς ε, πώς εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή και με ε, τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου. Θα πρέπει να είμαστε διαθέσιμοι και να συνεργαζόμαστε κατανοώντας καλά το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι δημόσιοι ελεγκτές και τι δεν μπορούν να κάνουν η βασική ευθύνη είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δώσει πληροφορίες για τους ε, λογαριασμούς, τα λογιστικά, ε, την κανονικότητα αυτών των λογιστικών και τα αποτελέσματα γενικότερα ρόλος του συνεδρίου είναι να παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες και κυρίως ανεξάρτητες εγγυήσει για τα προηγούμενα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής και όπως είπε και η κυρία Σέντερ να βοηθήσει το Κοινοβούλιο να αναζητήσει καλύτερη σχέση ε, κόστους και ωφέλους για τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλους τους τομείς των δαπανών. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Εμείς ελέγχουμε τα δημοσιονομικά, ελέγχουμε επίσης και το κατά πόσον είναι συμβατές οι λογιστικές ενέργειες που γίνονται με τα διεθνή λογιστικά standards. Και όλα αυτά μπορεί να συνδυαστούν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς τις αρμοδιότητες να κάνουμε εκ των υστέρων ε, λογιστικούς ελέγχους όλων των τριών ε, τύπων ε, λογιστικής διαχείρισης, τότε δεν θα έχουμε μια αξιόπιστη βάση έτσι ώστε να προειδοποιούμε και εσάς και τους πολίτες για τους κινδύνους τους οποίους δημιουργεί η ε, συγκεκριμένη μορφή οικονομικής διαχείρισης και να μην παρέχουμε επίσης και τους προσανατολισμούς τους οποίους ζητάτε και να βελτιώνουμε την οικονομική διαχείριση. Γι' αυτό ακριβώς το ελεγκτικό συνέδριο έχει εμπλακεί ήδη στην επεξεργασία ορισμένων θέσεων. Σας είχα ενημερώσει και για το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2013 στην αρχή του έτους. Ήδη έχουμε αρχίσει και καλύπτουμε κάποια από τα θέματα τα οποία υπογραμμίζει η έκθεση Σέντερ ε, για τις DAS. Προσπαθούμε εμείς να βελτιστοποιήσουμε το μέσο αυτό ε, για την αξιολόγηση της χρήσης των κοινωνικών, κοινοτικών πιστώσεων. Ε, η ομάδα εργασίας για τα λογιστικά και την οικονομική κρίση προσπαθεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει το θέμα της έκθεσης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική κρίση, αλλά και προσπαθεί να δει ποιες είναι πραγματικά οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του σχεδιασμού όλων των μηχανισμών εξόδου από τη συγκεκριμένη κρίση. Έχουμε επίσης και το θέμα της παραγωγής των ειδικών εκθέσεων προσπαθούμε να κάνουμε και τα λεγόμενα landscape reviews για τους κινδύνους τους οποίους εμπεριέχουν οι διάφορες λογιστικές μορφές ελέγχου. Είναι προς όφελος λοιπόν και του Κοινοβουλίου το συνέδριο να συνεχίσει να ε, ασκεί όλα τα δικαιώματα που έχει και για τους εκ των υστέρων εξ ελέγχους. Και όλα αυτά θα πρέπει βέβαια να συνοδεύονται και από τους πόρους που είναι απαραίτητοι και οι κανόνες εξάντε, εκ των προτέρων, σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους στο ε, χρηματοοικονομικό σύστημα. Μεγαλύτερη εμπλοκή όλων των ευρωπαϊκών οργάνων στον καθορισμό των προγραμμάτων και στον προγραμματισμό των ελέγχων όλα αυτά θα μπορούσαν εν μέρη να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία του συνεδρίου και την ικανότητά του σύνεπως να φέρει πέρα τον ρόλο, εις πέρα στον ρόλο του σαν ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο. Η συνθήκη εδώ είναι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργάζονται προς όφελος όλων. Και πιστεύω, Πρόεδρε, ότι η βασική αρχή της διοργανικής συνεργασίας θα πρέπει να προσανατολίζει και να καθοδηγεί την κοινή μας δράση αναζητώντας ε, την ε, καλύτερη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ένωση και τον πολίτη. Το συνέδριο λοιπόν είναι θεμελιώδες να παραμείνει ανεξάρτητο, επαγγελματικό και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο να έχει τους ιδίους στόχους με όλα τα άλλα όργανα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την κυρία Γιάλα Σέντερ για την ευκαιρία που μου δώσατε και θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω και τις πρώτες θέσεις του συνεδρίου σε γραπτή μορφή το ταχύτερο δυνατόν είμαι, ε, στη, θα είμαι στη διάθεσή σας τα επόμενα έτη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε Καλτέρα. Δύο μιλητές ήδη έχουν ζητήσει το λόγο. Γκερμπράντι ο πρώτος. Και ο επόμενος ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά εκ βάθους καρδίας την κυρία Γιάλα Σέντερ, διότι συμφωνώ απολύτως σε μεγάλο βαθμό με την έκθεσή ε, της. Δηλαδή, στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής, να, ε, όχι μόνο στο νομότυπο, να δίνει την έμφαση το ελεκτικό συνέδριο. Το 2009, όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά, εξεπλάγει που το ελεκτικό συνέδριο δεν έδινε τόση προσοχή σε αυτό. Ευτυχώς όλο και περισσότερο το πράττουν ε, και στις ειδικέ εκθέσεις προκειμένου. Επίσης, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο με την κριτική σας και τις επικρίσεις ε, ε, να υπάρχει ένα μέλος, ένα κράτος μέλος, ένα μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα πολύ μεγάλο αριθμό μελών ε, του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά θίγει και το ζήτημα της ανεξαρτησίας, που για μένα είναι το πιο σημαντικό στη λειτουργία του ελεκτικού συνεδρίου. Το στοιχείο της ανεξαρτησίας θα πρέπει να είναι δεδομένο και να ε, υπάρχουν τα εχέγγυα γι' αυτό. Ε, δεν συμφωνώ τόσο πολύ με την πρόταση της κυρίας Αγιάλα να αποφασίζουν και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το πολιετές πλαίσιο ε, και ε, τις επιλογές γιατί έτσι κάπως θίγεται η ανεξαρτησία. Και μπορεί να είναι και πολιτική επιλογή πάντα ε, η προτεραιότητα του καθενός. Καλά θα κάνουμε λοιπόν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να μην αγγίζουμε αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, εντάξει να κάνουμε προτάσεις αλλά να τους αφήνουμε να αποφασίζουν μόνοι τους. Για το Διοικητικό Συμβούλιο τώρα δεν μπορούμε να έχουμε εκπροσώπους και από τα 28 κράτη-μέλη. Νομίζω ότι στην πράξη αυτό δεν είναι πάρα πολύ ε, σκόπιμο ούτε λογικό. Το πιο σημαντικό για μένα ε, ως προς την ανεξαρτησία είναι το εξής. Ανησυχώ εγώ με την όλο και περισσότερη πολιτικοποίηση στο διορισμό των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Το είδαμε τα παρελθόντα έτσι με τον Ισπανό υποψήφιο, τον Ιρλανδό και τώρα δυστυχώς συμβαίνει το ίδιο και με τον Ολλανδό υποψήφιο. Ο κύριος Ντεφρίς είναι εξαιρετικό ε, πρόσωπο ε, και έχει και το ιδεώδες προφίλ για να είναι εκεί και τον αντικαθιστούν για λόγους πολιτικούς. Το θέμα δεν είναι ποιος θα τον αντικαταστήσει, αλλά δεν μπορεί κομματικά κριτήρια να ε, καταργούν ε, ένα εξαιρετικό μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό. Τέλος. Του Πρόεδρε. Ε, μιλούμε και για το ρόλο του ίδιου του Κοινοβουλίου. Τώρα εμεί έχουμε ένα απλό συμβουλευτικό ρόλο ε, κατά το διορισμό των μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Είδαμε με τον Κροάτι υποψήφιο πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό. Εγώ ε, θα παραμείνω στην άποψή μου και θα ζητήσω να έχουμε και ρόλο αποφασιστικό, όχι μόνο συμβουλευτικό. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι προς την κατεύθυνση αυτή. Και μια τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε. όλο και περισσότερο με ενοχλεί ότι δεν δίνεται μεγάλη συνέχεια στις γνωμοδοτήσεις, στις συμβουλές ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Το ξέρω ότι είναι περίπλοκη ευρωπαϊκή νομοθεσία από τον χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό κανονισμό. Όλο και περισσότερο μας λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι αυτή η περιπλοκότητα είναι εμπόδιο ε, και ούτε η Κομισιόν, ούτε το Συμβούλιο, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούνε αρκετά όσα λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Και επίσης μας λένε ότι δεν είναι αποτελεσματικά αυτά που κάνουμε. Για το αγροπεριβαλλοντικό ας πούμε πρόγραμμα που χρόνο με το χρόνο λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι με αυτά τα μέσα που έχουμε δεν φτάνουμε στο στόχο μας. Δεν υπάρχει δηλαδή σχέση αιτίου και αιτιατού με τους πόρους που διαθέτουμε σε ένα στόχο αύριο, μάλλον σήμερα το πρωί, ε, απερίφθη η τροπολογία μου στην Επιτροπή Προπολογισμού. Κρίμα το 10% της πίστοσης να μπει στο αποθεματικό για να δείξουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, δεν επιτυχάνονται οι στόχοι με σωστό τρόπο. Τώρα θα μπορούσα να κάνω ξεχωριστή συζήτηση ε, ολόκληρη για το τι μοίρα επιφυλάσσουμε ε, στις γνωμοδοτήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου δεν αφορά μόνο το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάντως, είναι εξαιρετική έκθεση κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ κύριο Ζαμπιεροντή. Euh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την αποφασιστικότητα, την αφοσίευση της συναδέλφου Αγιάλα Σέντερ πάνω στο θέμα αυτό να πω ότι έχουμε μια καλή συζήτηση μεταξύ μας για να ορίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε μια κάποια δυσφορία η οποία υπάρχει γύρω από το θέμα του δημοσιονομικού ελέγχου στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων. Είναι σαφές ότι έχουμε μια συλλογική συνευθύνη ε, και σε επίπεδο κοινοβουλίων, κυβερνήσεων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι και το αντικείμενο. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορέσουμε να πούμε τα πράγματα με ξεκάθαρο τρόπο. Θα ήθελα να υποστηρίξω την πρόταση λοιπόν του κυρίου Καλτέρα. Όχι να υποστηρίξω, αλλά πώς να σας το πω. Να ωφεληθώ από την πρόταση του να μας δώσει τη γραπτή άποψη του ε, συνεδρίου στις συζητήσεις μας πριν χωρίσουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι τις θέσεις ε, των παρέδρων του συνεδρίου ε, στα πλαίσια της διαμόρφωσης των θέσεών μας. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά πάντως θα υποστηρίξω την ιδέα η οποία ακούγεται να μπορέσουμε το έγγραφο του συνεδρίου να το εντάξουμε στις συζητήσεις μας. Τώρα για τις προτάσεις γενικότερα, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε όλοι σαν βασικό στόχο τον σεβασμό των λεγόμενων διεθνών κανόνων. Δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε τον κανόνων αυτών. Γιατί αλλιώς θα φανούμε σαν κάποια μορφή ιδιορυθμίας αυτοδιαχειριζόμενης. Όχι, οι διεθνώς ισχύοντες κανόνες και η λογιστική που δεν είναι το θέμα μας αλλά η ελεγκτική που ορίζονται από τους δημοσιονομικούς ελεγκτές είναι αυτοί που θα πρέπει να ισχύουν. Τι λέγουν οι κανόνες αυτοί. Λέγουν ότι τα ανώτατα Ινστιτούτα ελέγχου, τα ανώτατα όργανα ελέγχου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και είμαι πολύ επιφυλακτικός με την ιδέα που ακούστηκε το ελεγκτικό συνέδριο να βασιστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την χορήγηση των βεβαιώσεων DAS. Ίσως εδώ να υπάρχει ένα θέμα περαιτέρω ανταλλαγής απόψεων. Πάντως, η συνεργασία ανάμεσα στον εσωτερικό έλεγχο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εξωτερικό που κάνει το συνέδριο καθορίζονται σε επίπεδο διεθνούς νομοθεσίας. Εκεί θα βρούμε πολλά πράγματα για να κάνει περισσότερα το ελεγκτικό συνέδριο σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ανεξάρτητη. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής δεν είναι ανεξάρτητοι και δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο που θα οδηγήσει στη χορήγηση των DAS. Δεν ισχύει το ίδιο για τις ανώτατες ελεγκτικές εθνικές υπηρεσίες. Εγώ είχα πει ότι τα πιστοποιητικά αυτά, τα DAS για τα δημοσιονομικά μπορούν να γίνουν μέσα από ελέγχους των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων και στα πλαίσια του εγγράφου για τη μεθοδολογία των DAS, των δηλώσεων αξιοπιστίας, ε, είναι σαφές ε, ο, ο λόγος, είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ε, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια είναι ανεξάρτητα. Αυτό δεν ισχύει για τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης και στην αλυσίδα των εσωτερικών ελέγχων έχουμε τον ρόλο και των δημοσίων υπηρεσιών. Είχα πάει στην Γαλλία μαζί με την Κρέσλε ε, είδα τον διευθυντή, είδα τους, τις αμοιβέ του, τον τρόπο με τον οποίο διορίζεται. Είμαι πεπισμένος ότι ο υπάλληλος αυτός ελέγχεται από τον Υπουργό και δεν είναι ανεξάρτητος ελεγκτής, ενώ το ανώτατο ελεγκτικό συνέδριο της κάθε χώρας είναι ανεξάρτητο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα για τα προγράμματα εργασίας, στην παράγραφο 12 θα πρέπει να λάβει υπόψη το συνέδριο τους ρυθμούς εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνεισφέρει σε αυτούς. Πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει μια κάποια διαβούλευση, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στον καθορισμό του δικού του προγράμματο εργασίας που είναι θέμα πολιτικό και όχι τόσο θέμα εκ ε, ε, ελέγχου. Το ίδιο αισθάνομαι επίσης και για την παράγραφο 15 ότι δηλαδή το συνέδριο θα μπορούσε να παρέμβει στις νομοθετικές προτάσεις ε, του συνεδρίου. Έχω την αίσθηση ότι σε κάθε δημοκρατία υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο καταρχάς αυτό το οποίο κάνει είναι ο πολιτικός έλεγχος και ο δημοσιονομικός έλεγχος και ο έλεγχος του εκτελεστικού. Και εδώ ακριβώς το ελεγκτικό συνέδριο παρέχει μία γνωμοδότηση στον ελεγκτή που είναι το κοινοβούλιο. Συνεπώς θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε όλα αυτά αρκετά καλύτερα ακόμα Πάντως είμαι πεπισμένος για την ανάγκη μιας ανεξάρτητης μορφής ελεγκτικού συνεδρίου και μιας δήλωσης, μιας δήλωσης αξιοπιστίας, μιας ντάσης η οποία να είναι συμβατή και αναγνώσιμη. Η, τα λογιστικά είναι εγκεκριμένα εν πάση περιπτώσει ναι ή όχι. Οι συστάσεις που είχαν δοθεί εφαρμόστηκαν ναι ή όχι και αυτό το οποίο θα κάνω είναι να προτείνω τροπολογίες γιατί όταν τα ντάς, όταν οι δηλώσεις αυτές δεν ε, έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Βρισκόμαστε σε μια μυστήρια κατάσταση όπου δεν υπάρχει κύρωση όταν υπάρχει αρνητική ντάς. Όταν υπάρχει μια αρνητική τέτοια δήλωση θα πρέπει το Κοινοβούλιο να προχωρά σε βέτο ακόμα αν θέλετε και της Επιτροπής και να υπάρχουν κυρώσεις. Εγώ όπως σας είπα έχασα τροπολογίες για το GNSS όπου είχα πει ότι όταν ένας εκτελεστικός διευθυντής έχει αρνητική απαλλαγή θα πρέπει να υποβάλει την παρέτησή του. Δεν έγινε δεκτή η πρότασή μου, θα επανέλθω όμως. Δεν μπορεί να υπάρχει μια αρνητική απαλλαγή σε μια υπηρεσία και ο εκτελεστικός διευθυντής στο διοικητικό συμβούλιο να συνεχίσουν σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι θα έλεγα η προσπάθεια έλλειψης αξιοπιστίας της ίδιας της ελεγκτικής διαδικασίας. Τώρα, για την οργάνωση την θεσμική και για τη δυνατότητα ενός διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα καταστήσει το ελεγκτικό συνέδριο σαν μια ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία. Ε, διαφωνώ. Η σημερινή οργάνωση με μέλη του συνεδρίου ανεξάρτητα. Νομίζω ότι αυτού του τύπου η δομή είναι καλή και δεν πρέπει να προσαρμοστεί σε μια άλλη μορφή λειτουργίας μέσω, ελεγκτικού, μέσω ε, διοικητικού συμβουλίου. Τώρα και για τους τρόπους ορισμού των μελών θα συμφωνήσω με την συνάδελφο Γιάλα Σέντερ. Εξέφρασα τη λύπη μου για αυτά τα οποία είχαν συμβεί με τον Ισπανό υποψήφιο. Η πολιτική μου άδα με είχε επιφορτήσει ε, με τον ρόλο του σκιώδου εισηγητή στο θέμα του ορισμού. Με λυπάται η Νομίζω εν πάση περιπτώσει ότι το πρόσωπο που θα ορίσει τον ελεγκτή να είναι αυτός ο οποίος θα εγκρίνει τις υπηρεσίες του σε μία, στο ιδιωτικό επίπεδο. Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον ελεγκτή και οι συνθήκες αμοιβή του είναι τέτοιες έτσι ώστε να παραμένει ανεξάρτητος. Τώρα, σήμερα, οι κυβερνήσεις ε, ορίζουν, διορίζουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Αποσύρουν ε, εναντίον άλλωστε συχνά και της άποψης του Κοινοβουλίου κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του ελεγκτικού, της ελεγκτικής διαδικασίας. Οι συνάδελφοι στα Εθνικά Κοινοβούλια ελέγχουν τα εθνικά εκτελεστικά όργανα θα πρέπει να δεχτούν κάποιες προτάσεις, αλλά θα πρέπει πρώτα το Κοινοβούλιο ε, να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία ορισμού των ελεγκτών. Τώρα μετά από πρόταση των κυβερνήσεων αυτό δεν είναι κακή διαδικασία και αυτό το συμβούλιο που προβλέπεται στο σύνολό του, το συμβούλιο μάλλον ε, υπουργών συνολικά να μπορεί να βάζει ένα είδος βέτο έτσι ώστε ε, να προλαμβάνονται καταστάσεις περιθωριακές που μπορεί να προκληθούν από τον ε, καταμερισμό των πολιτικών δυνάμεων σε ένα κοινοβούλιο. Αλλά μία κυβέρνηση και το είδαμε στην κροατική περίπτωση μετά από μία ψηφοφορία να επιβάλλει έναν ε, ελεγκτή, ένα μέλος του συνεδρίου, αυτό είναι απαράδεκτο. Το Κοινοβούλιο είναι ο πρώτος βασικός χρήστης των υπηρεσιών του ελεγκτικού συνεδρίου, πρέπει να συμμετέχει στον ορισμό και στη σύνθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις συνθήκες. Λοιπόν αυτά είχα να σας πω. Να πω για μια ακόμη φορά ε, στη συνάδελφό μου ότι είμαι επιφυλακτικός για κάποιες από τις προτάσεις της, αλλά θέλω να την ευχαριστήσω για τις ακροάσεις που διοργάνωσε, για τα θέματα που έθεσε και για τις προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν για να ξεφύγουμε από αυτή τη δυσθυμία, από αυτή τη δυσφορία που επικρατεί σε ό,τι έχει σχέση με ε, τον έλεγχο και τις ελεγκτικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Καλά λοιπόν, αφού δεν επιθυμεί κανείς άλλος. Τότε, πριν να ζητήσω, πριν να παρακαλέσω την ε, κυρία Γιάλα Σέντερ να λάβει τελευταία το λόγο, κύριε Οντή, μιλήσατε για το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 17 Δεκάτου Οκτωβρίου. Το μεσημέρι. Αν ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από τον κύριο Καλντέρα, τίθεται ερώτημα, κρατούμε αυτή την ημερομηνία. Για την ώρα, ας το δουν οι συντονιστές μας. Αν βρουν κάτι που για αυτούς έχει κρίσιμη σημασία, Ίσως η κυρία Γκρέσλε και οι συναδελφοί της, ο κ. Σκάιερ, να προτείνουν ενδεχομένως παράταση κατά ένα μήνα. Μετά, 7 Νοεμβρίου, έχουμε προβλέψει την τελική ψηφοφορία, ώστε να προχωρήσει η ε, έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Θα είμαστε λοιπόν εύκαμπτοι σε ό,τι αφορά την ε, παράταση της προθεσμίας, αλλά μόνο εφόσον ε, δούμε ότι είναι πραγματικά απαραίτητο. Τώρα. Ίσως μπορούμε να προβλέψουμε κάποια απαγόρευση ε, να ε, προτείνεται από κάποια πλειοψηφία, κάποιος εθνικός ε, αντιπρόσωπος στο ελεγκτικό συνέδριο. Εσείς ε, όμως κύριε Οντή νομίζω θέλετε να παρέμβετε και πάλι για λίγο. Ναι, σύντομα για το χρονοδιάγραμμα. Το έγγραφο του κυρίου Καλντέρα, Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα είναι σημαντικό διότι θα μας μεταφέρει τις απόψεις του συνεδρίου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η έκθεση να καταλήξει την Ολομέλεια πριν να αρχίσει η προεκλογική εκστρατεία, διότι το θέμα αυτό ενδέχεται να πέσει στα χέρια των πολιτικών κομμάτων. Α τα ακούσει αυτά και η συγκήτρια και να υποβάλει τι ε, τροπολογίε τη ενδεχομένω στην Ολομέλεια. Να μην παραταθεί δηλαδή υπερβολικά το χρονοδιάγραμμα, διότι πρέπει όντω να έχει τελειώσει, να έχει ψηφιστεί τελικά δηλαδή ε, η έκθεση πριν από τι εκλογέ. Ο κύριο και ευχαριστώ. Εσεί αγαπητοί παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλτέρα, βέβαια έχει ήδη αποχωρήσει. Ε, τον ευχαριστώ για ε, τον κόπο του που ήρθε. Το ξέρω, τον ενδιαφέρε και τον ίδιο. Σημειώνω τις ανησυχίες των συναδέλφων και τα μελήματά τους. Είναι γεγονός ότι το είχα πει και εγώ, ένα ανεξάρτητο ελεγκτικό συνέδριο είναι και για μένα σημαντικό όσο και για τους άλλους. Αλλά επίσης σημαντικό είναι να μετράει και η γνώμη του. Και να έχει νόημα να εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Μου έχει συμβεί και εμένα. Και για τώρα λόγο μέλος του, του ελεγκτικού συνεδρίου να έχει έρθει η ε, γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου ενώ το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, δαπανηθεί, ε, διεκπαιρεωθεί και ξεχαστεί. Δηλαδή, λέμε εκ των υστέρων, αλλά είναι τόσο εκ των υστέρων που είναι πραγματικά μετά το τέλος. Και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δουλειά που έχουν προβλεφθεί ε, τι νομοδοτήσει. Καλή ανεξαρτησία. Αλλά θα πρέπει να έχει νόημα. Δεν ξέρω πώς θα η διατύπωση. Δεν εννοούσα αυτό που καταλάβατε. Δεν θέλω το ελεγκτικό συνέδριο να είναι ένα ε, μέσον το οποίο να βαρύνει μόνο εκ των υστέρων και εκ των προτέρων να έχει λόγο. Γιατί παίρνονται αποφάσεις στο Συμβούλιο, στο πόδι, για να μην πω νυχτιάτικα, που καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, και έχουν επιπτώσεις και για τον κοινοτικό προπολογισμό και για τους κρατικούς προϋπολογισμούς χωρίς να συμμετέχει καθόλου ε, προληπτικά, αν θέλετε, το ελεκτικό συνέδριο. Είναι και δική τους ε, αγωνία αυτό. Δεν θέλουμε πάντα να είναι επιμηθείς. Να είναι και προμηθείς καμιά φορά το ελεκτικό συνέδριο. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αμφισβητήσω την ανεξαρτησία του ελεκτικού συνεδρίου αλλά να έχουν νόημα, να μην έρχονται οι άνθρωποι να γνωμοδοτούν και μετά να μην λαμβάνεται υπόψη, να είναι πολύ αργά, να μην χρησιμεύουν σε τίποτα οι γνωμοδοτήσει. Να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, τι άλλο. Για τη σύνθεση του, συμφωνώ με κάποιες από τις επικρίσεις που ακούστηκαν, αλλά επίσης θα ήθελα να μπορούμε να συζητήσουμε, στις τροπολογίες θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, για τις δυνατότητες που έχουμε έτσι ώστε να βελτιώνεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τρόπο διορισμού των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Γιατί να δίνουμε απλούστατα την ικανοποίηση στο Συμβούλιο να απορρίπτει τη δική μας πρόταση. Δεν μου αρέσει αυτό, γιατί εμείς όταν έχουμε μια απορριπτική εισήγηση να ισχύει αυτό και όχι να μας αγνοεί το Συμβούλιο. Αυτά. Για το χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, δεν θέλω η έκθεσή μου κάπου να τοποθετηθεί και να ξεχαστεί παρκαρισμένη, γιατί το καινούριο κοινοβούλιο δεν ξέρω και τι προτεραιότητα θα της δώσει και πόσο θα το ενδιαφέρει. Το είπε και ο κύριος Σοντή, θα μπορούσαμε και στη συζήτηση τη δική μας στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια να έχουμε και τις ιδέες του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά να μην φρενάρουμε το χρονοδιάγραμμα μας σε τρόπο που να είναι επικίνδυνος, αλλά να έχουν τη δυνατότητα και εκεί να εκφραστούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. At this moment, let us close the item. Ας ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση του θέματος 8 και ας προχωρήσουμε, ας επιστρέψουμε στο 7, όπως αρχικά είχε ε, προταθεί. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πίπερ, λοιπόν, μετά στον Επίτροπο Σέμετα και μετά στην κυρία Καριουλάιτη πάλι του, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κύριε Πίπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να κάνω μια σύντομη εισαγωγή και πρώτα επιθυμώ να ευχαριστήσω ρητά την Επιτροπή, τον Επίτροπο κύριο Σέμετα για την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, την οποία είχε ούτως ή άλλως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία έκθεση με τη μορφή που έχει υποβληθεί τώρα και το λέω αυτό με πεποίθηση αποτελεί πραγματικό στήριγμα για μας ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια ε, δημοσιονομικές διορθώσεις και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην ε, αξιολόγηση του σφάλματος, του ποσοστού σφάλματος στις διάφορες χώρες μέλη. Βέβαια, ασφαλώς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να ζητάμε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάντως για την έκθεση που βάλατε κύριε Επίτροπε και καταρχήν θα πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Πριν τώρα ε, κάνετε την παρέμβασή σας, επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, ίσως μάλιστα να προσθέσω και ορισμένες ερωτήσεις που μπορείτε μετά να απαντήσετε. Κάτι που επισημαίνω είναι ότι υπάρχουν ορισμένες λίγες χώρες μέλη οι οποίες αφορώνται από τις δημοσιονομικές διορθώσεις του 2012 αλλά λίγε χώρες είναι εκείνες οι οποίες είναι υπεύθυνε για το 70% των σφαλμάτων. Έχουμε και μια χώρα και δεν πίστευα τα μάτια μου, την Ισπανία, η οποία φέρει την ευθύνη για 58% των ανακτήσεων. Και μάλιστα άλλη μια φορά δεν πίστεψα ε, τα μάτια μου με το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο συνολικά 2.416 υποθέσεις και από αυτές περίπου 900 στην Ισπανία. Τι να πω. Ως βουλευτής έχω μείνει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Πώς είναι δυνατόν. Παρακαλώ να μου δοθεί πρώτα μια εξήγηση από πλευράς Κομισιόν. Πριν να προβληθούν και άλλες αξιώσει από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, για διευκρίνηση δηλαδή, αν είναι δυνατόν κάποια πράγματα από αυτά να διευκρινίσετε. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα ή περιφέρειες οι οποίε βρίσκονται σε βαθιά κρίση να πηγαίνουν τα πράγματα τόσο άσχημα και στις δημόσιες ε, προμήθειες. Ίσως έκλεισαν κάπου ένα μάτι, ίσως έκλεισαν και τα δύο μάτια έτσι ώστε να κρατήσουν τα λεφτά στην περιφέρειά τους. Αυτό ίσως αποτελεί μια εξήγηση, ίσως, όχι βεβαίως δικαιολογία. Γιατί εν τέλει, εάν δεν έχουν γίνει νομότυπα οι διαδικασίες αυτές, βλάπτεται τελικά η ίδια η περιφέρεια. Με ενδιαφέρει λοιπόν να δω πώς κρίνεται, εκτός από την Ισπανία είναι και η Ελλάδα και η Ιταλία. Και πιθανώς θα προσθεθεί και η Πολωνία αλλά και η Ρουμανία. Πώς λοιπόν μπορείτε να εξηγήσετε την κατάσταση αυτή που συμβαίνεται σε αυτές τις χώρες. Ποιες είναι οι αιτίες, καθώς επίσης ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία συνάγεται. Διότι μπορείτε να είστε βέβαιος ότι πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες δεν λαμβάνουμε μόνο εμείς εδώ της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Είναι πια δημόσιο κτήμα και θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από πλευρές που δεν είναι τόσο ας πούμε φιλοευρωπαϊκές και εάν δοθούν από εσά κάποιες πιστικές απαντήσεις να δούμε τέλος πάντων που, προς τα που θα προχωρήσουμε. Θα δείξω αυτοσυγκράτηση πάντως εν προκειμένου Έχουμε ήδη προβληματιστεί σχετικά με το ποιε απαιτήσει μπορούμε να προβάλλουμε από πλευρά Κοινοβουλίου, αλλά θα μου δοθεί και πάλι ο λόγο μετά. Γι' αυτό θα υποβάλω μετά και άλλε ερωτήσει. Για παράδειγμα, αυτέ οι ακραίε διαφορέ μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερική Ανάπτυξης, όπου στο Κοινωνικό Ταμείο έχουμε ποσοστά ανακτήσεων 91% και στο άλλο ταμείο 28,8% δηλαδή το Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως. Πρόκειται για τεράστιες διαφορές. Πώς μπορούν να εξηγηθούν. Και μία παρατήρηση ακόμη για αυτή τη λεγόμενη επιχρήσωση. Δηλαδή αυτούς τους κανόνες που έχουν κάνει ακόμα περιπλοκότερους οι χώρες μέλη. Είχαμε και μια καλή έκθεση του Γιένς Γκάιερ και είχαμε ζητήσει να μας δοθούν απαντήσεις γιατί και σε ποιο βαθμό οι χώρες μέλη επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις και ποιες ποια μπορεί, ποια μπορεί να είναι τα συμπεράσματα. Εσείς δυστυχώς επαναλάβατε τις απαντήσεις σας του προηγούμενου έτους. Ουδέν νέο στοιχείο, παρόλο που η κατάσταση περιγράφηκε καθαρά από τον κύριο ε, Γκάιερ. Δηλαδή η υπόθεση αυτή του gold plating της επιχρήσωσης δεν έχει απαντηθεί κατά την κρίση μας επαρκώς. Αυτά ως μια πρώτη τοποθέτηση. Στην πρώτη μου αυτή λοιπόν τοποθέτηση θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτή την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων, κάτι που βλέπω να λείπει, εφόσον μιλάτε για προστασία του προϋπολογισμού, πού υπέστη βλάβη ο προϋπολογισμός, σε ποιο βαθμό μπορούμε να πούμε ενδεχομένως με διαφυγή εσόδων από τόκους, από καθυστερήσεις διαδικασιών σε χώρες μέλη διότι χάνονται χρήματα, χάνεται πραγματικό χρήμα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει και ένα βήμα ακόμα έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθούν οι συνέπειες αυτών των σφαλμάτων και οι καθυστερήσεις της ανακτήσεις για παράδειγμα. Διότι αυτό θα συνιστούσε μια ακόμα ειλικρινέστερη απάντηση για τέτοια πράγματα τα οποία εξοργίζουν. Δεν θα ολοκληρώσω ωστόσο χωρίς να πω ότι χαρήκαμε κιόλας διότι σε 22 χώρες μέλη προφανώς τα πράγματα λειτουργούν. Δηλαδή τα ποσοστά σφαλμάτων ή οι διαδικασίες ανακτήσεων ανέρχονται στο 3,5% και για μεγάλα χρονικά διαστήματα τώρα έχουν γίνει αυτοί οι υπολογισμοί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι διαδικασίες κυρώσεων, ανακτήσεων, επιθωρήσεων, ελέγχων και της Κομισιόν αλλά και των χωρών μελών φαίνεται να έχουν κάποια απόδοση. Και τέλος θέλω να ρωτήσω, τι θα κάνουμε τώρα με τους λίγους κακούς μαθητές, ποιες συστάσεις, ποια συμπεράσματα εξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτή την εσφαλμένη, την κακή συμπεριφορά ορισμένων χωρών μελών. Α, και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, μία ακόμη παρατήρηση. Το ερώτημα απευθύνεται όχι μόνο στην Κομισιόν, αλλά βεβαίως και στο ελεγκτικό συνέδριο. Γνωρίζω ότι και ε, το, και το όργανο αυτό προβληματίζεται τι θα γίνει με αυτούς τους ε, παράτυπους και ενδιαφέρομαι, αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Γνωρίζω ότι η κυρία Αργιουλάιτε είναι παρούσα. Κύριε Πίπερ, σας ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά δίνω το λόγο τώρα στον Επίτροπο κύριο Σέμετα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή σας για τα εισαγωγικά του λόγια. Πρόθεσή μου ήταν να παρουσιάσω τρεις εκθέσεις που συζητούνται και εδώ στο σώμα αλλά και τις προοπτικές για την ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων που αναφέρατε και εσείς στην τοποθέτησή σας. Ας αρχίσω με την σύνθεση report και πρώτα να τονίσω ότι αυτό το σημαντικό έργο λογοδοσίας είναι αποτέλεσμα των προσπάθειών μας και αυτά προκύπτουν από τις εκθέσεις, τις εκθέσεις δραστηριότητων. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι οι εκθέσεις δραστηριοτήτων προβαίνουν σε αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 15 γενικοί διευθυντές και δύο διευθυντές οργανισμών έχουν προβάλει 29 συνολικά επιφυλάξεις. Τα συνολικά ποσά είναι μεταξύ 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μεταξύ 1,9 και 2,6% όλων των εκτελεστισών πληρωμών. Ταυτόχρονα οι δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά και φτάνουν στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ του 2011. Θα εξηγήσω σε λίγο ότι αυτή η αξιολόγηση αποδίδει σωστά την δημοσιονομική έκθεση των τελευταίων ετών. Η σύνθεση report περιλαμβάνει τώρα και συγκεκριμένες οδηγίες προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ιδίως για τα εξής ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων των διαδικασιών προμηθειών. Επίσης, κριτήρια υλοποίησης που είναι σημαντικά για την αύξηση της συνέπειας και συνεκτικότητας των οργάνων αξιολόγησης, επιλογές, κόστους για την αντικατάσταση ορισμένων εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που είναι δυσκίνητη, επίσης για διακοπή και αναστολή πληρωμών, για το 2012 για την πολιτική συνοχής 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ διακόπηκαν ως πληρωμές και αναστάθηκαν τέσσερα προγράμματα στην Ιταλία, Γερμανία, Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακική Δημοκρατία. Η ενεργός εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων οδήγησε σε σημαντική αύξηση των ποσών που αποκλείστηκαν από τις τακτικές πληρωμές, όπως θα εξηγήσω και στην για την έκθεση για την προστασία του ε, προϋπολογισμού της Ένωσης. Τώρα, οι νέες ε, διατάξεις ενισχύουν τις ε, υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης των χωρών μελών και η Κομισιόν ενθαρρύνει την χρήση εθνικών δηλώσεων όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το νέο πλαίσιο. Οργανώνω μαζί με τον Γιάνν Μιούλντερ μια ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό, ώστε να προταθεί ένα συνολικό, ένα κοινό template που θα αρχίσει να λειτουργεί από του χρόνου. Τέλος, η Κομισιόν προωθεί σε όλες τις, τις υπηρεσίες μια νέα νοοτροπία που θα εφαρμόζει στη νέα γενιά προγραμμάτων την δημοσιονομική προοπτική των ετών 2014-2020. Τέλος, όσον αφορά την έκθεση αξιολόγησης της του άρθρου 319 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη, σας, υπόψη της τις τις σας για βελτιώσεις. Όσον αφορά δε το χρονοδιάγραμμα, η Κομισιόν ήδη ενέκρινε σχετική έκθεση τον Ιούνιο φέτος. Όλοι οι τομείς πολιτικής καλύπτονται και οι συμβολές των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 περιλαμβάνονται όπου υπάρχει τέτοια πληροφορήση. Η, η σύνθεση report βασίζεται στη συμβολή διαφόρων υπηρεσιών της Επιτροπής και μεταξύ αυτών και των ελεγκτών που περιλαμβάνει τις πιο, σημαντικές, τα πιο σημαντικά συμπεράσματα των ελέγχων και από τις υπηρεσίες κομισιών και από τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Μεταξύ των 29 auditing engagements του 2011 να σας μιλήσω για δύο οριζόντιους ελέγχους που δείχνουν πώς γενικά βελτιώνεται η διαχείριση από πλευράς Κομισιόν και η ενημέρωση. Πρώτα, ο έλεγχος για την διαδικασία ετησίων εκθέσεων, ο εσωτερικός έλεγχος βρήκε ότι η διαδικασία λειτουργεί καλά, αλλά χρειάζεται και άλλες βελτιώσεις, ιδιαίτερα εκθέσεις για την ορθή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δομή των εκθέσεων ώστε να βελτιωθούν διαδικασία ποιότητας ελέγχων από πλευράς κεντρικών υπηρεσιών της Κομισιόν για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών. Αυτές οι βελτιώσεις θα είναι εφαρμοστές από το 2013 και μετά. Δεύτερο, για τα επιδόματα προσωπικού, για την σχετική παρακολούθηση, για να ε, ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπινων πόρων. Μεγαλύτερη λοιπόν διαφάνεια στην χρήση των πόρων, αναλόγως με τις προτεραιότητες και πιο αποτελεσματική ταυτοποίηση των αναγκών εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Τελειώνω τονίζοντας ότι σύμφωνα με την προτεραιότητα που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καθιέρωση μιας νέας νοοτροπίας κουλτούρας, δηλαδή της απόδοσης, οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούν μέχρι και 50% των πόρων τους για την αύξηση της αποδοτικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εντοπίσει ορισμένα από τα θέματα αυτά στα πλαίσια της απαλλαγής του 2011. Γι' αυτό και υποβάλλοντας την έκθεση για τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις της απαλλαγής, θα έλθω κυρίως στην πρόοδο που έχει γίνει σχετικά με τις τέσσερις δράσεις προτεραιότητας που έχετε περιλάβει στο ψήφισμά σας. Η πρώτη σας σύσταση ζητούσε από την Κομισιόν να συντάξει ανακοίνωση για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η ανακοίνωση, την οποία θα σας αναπτύξω αργότερα, καταδεικνύει ότι παρόλο που οι χώρες μέλη και οι Κομισιόν δεν μπορούν να προλάβουν όλα τα επιμέρους φάλματα, ωστόσο τα διορθωτικά μα συστήματα ε, προστατεύουν επαρκώ μακροπρόθεσμα τον κοινοτικό προπολογισμό. Επίση, η Κομισιόν έχει σημειώσει πρόοδο ό,τι αφορά την δεύτερη προτεραιότητα δράσεω που έχει σχέση με το ποσοστό σφαλμάτων. Ορισμένες από τι δράσει μα είναι οι εξή. Οι πρακτικές σχετικά με την διακοπή και αναστολή πληρωμών στι χώρε μέλη χρησιμοποιήθηκε εντατικά και όπου ήταν αυτό δυνατό εναρμονίστηκε. Οι διαδικασίες ελέγχων και δημοσιονομικών διορθώσεων επιταχύνθηκε. Λαμβάνουμε λοιπόν ε, φροντίδα ώστε να χρησιμοποιούμε πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και με μειωμένο κόστος. Όσον αφορά τη γεωργία, η Κομισιόν ενέκυψε στις ρίζες των σφαλμάτων στην εφαρμογή των ε, πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου. Ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ιταλία ήδη έχουν τροποποιήσει τα προγράμματά τους ανάπτυξη της υπαίθρου ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σφαλμάτων και για τη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπεται περαιτέρω εναρμόνιση των μηχανισμών διακοπής και αναστολής των πληρωμών στην πρόταση της Κομισιόν. Όπως εξήγησα και προηγουμένως η Κομισιόν δεσμεύεται για την εφαρμογή της τρίτης συστάσεως δράσεως της δικής σας, για τη βελτίωση δηλαδή των εκθέσεων αξιολόγησης και αυξημένη χρήση των ε, ελέγχων απόδοσης. Για τη νέα γενιά προγραμμάτων θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες, περιλαμβάνοντας στοιχεία που θα προσφέρουν ένα ισχυρότερο πλαίσιο απόδοσης, όπως με ευφυείς στόχους, καθώς και σχετικούς δείκτες, που θα βασίζονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα για την επίτευξη των στόχων προτεραιότητα της Ευρώπης 2020. Σε ό,τι αφορά την τέταρτη σύσταση για δράση για τους παραδοσιακούς ιδιού πόρους και τα έσοδα, έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη αφοροαποφυγή. Όσον αφορά τώρα του ε, δασμού και εκεί η Κομισιόν προωθεί αγώνα κατά της απάτης, με ε, ποινικέ διαδικασίες. Ήδη από το 2011 και μάλιστα έχει εγκρίνει και ανακοίνωση προ Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την εντατικοποίηση του αγώνα κατά του λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Το υψηλό επίπεδο εφαρμογής των συστάσεων του Κοινοβουλίου δείχνει ότι μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού και για τη χρηστή διαχείριση και ότι η Κομισιόν δεσμεύεται να αποδώσει. Κύριε Πρόεδρε, τέλος η πρώτη ανακοίνωση για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού, επί του οποίου ε, συγκεντρώθηκε ιδίω ο κύριος Πίπερ στην εισαγωγή του. Η προτεραιότητα της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι βεβαίω να προστίθεται αξία στους στόχους της Ένωσης. Η Κομισιόν όμως φέρει επίσης την ευθύνη μαζί και με τους άλλους ε, φορείς να προστατεύει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Για το λόγο αυτό, οι δράσεις που εφαρμόζονται για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιθεώρησης και ελέγχου της Κομισιόν. Η ανακοίνωση καθώς και τα παρατήματά της έχουν ως στόχο να δώσουν μια συνολική επισκόπηση του νομικού και οργανωτικού πλαισίου και να δείξουν τα αυτά αποτελέσματα των διορθωτικών δράσεων επί του προϋπολογισμού στο σύνολό του και ιδίως βέβαια στον τομέα των δαπανών. Τώρα έχω τα εξής νέα στοιχεία. Πρώτο, τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων ακολουθούν την αύξηση των πληρωμών. Για το 2012 δηλαδή έχουμε φτάσει στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 3,2% των πληρωμών που έγιναν. Λόγω του πολιετούς χαρακτήρα των ε, κοινοτικών δαπανών, οι δημοσιονομικές διορθώσεις γίνονται τα χρόνια μετά από το χρόνο που έγιναν οι πληρωμές. Οι διορθώσεις που έγιναν το 2012 αναφέρονται σε σφάλματα προηγουμένων ετών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου δεν είναι αποτελεσματικά για να ε, προστατεύουν διαρκώς τον προϋπολογισμό. Δεύτερο λοιπόν τώρα θέμα, η ειδική πληροφορία για την σύνδεση μεταξύ δαπανών και διορθώσεων σε ορίζοντα πλειώνων ετών έχει σχέση με, ε, να καταδείξει δηλαδή την ευρύτητα των μέτρων αυτών. Το σύνολο των διορθώσεων και ανακτήσεων για το 2009 έως 2012 ανέρχεται σε 2% του συνολικού όγκου των πληρωμών για την ίδια περίοδο. Ακόμα κι αν οι διορθώσεις αναφέρονται κυρίως σε πληρωμές που έχουν γίνει σε προηγούμενα έτη, το σχετικό εύρος των επιπτώσεων είναι και ένας δείκτης ότι λαμβάνονται υπόψη μαζί με τον δείκτη του ε, ποσοστού σφάλματος που έχει λάβει υπόψη του και το ελεγκτικό συνέδριο για τα έτη 2009 έως 2011. 3,3, 3,7 και 3,9%. Αν κοιτάξουμε ακόμη πιο πίσω, θα παρατηρήσουμε ότι από το 1994 με την κοινή διαχείριση παραπάνω από 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν γίνει αντικείμενο διόρθωσης, οριστικής διόρθωσης και οι διορθώσεις έχουν περιλάβει και άλλα 2 δισεκατομμύρια και εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τώρα τα ταμεία περιφερειακό και συνοχής για την περίοδο 2000-2006 που μπαίνει τώρα στην τελική φάση ο έλεγχος δηλαδή ανέρχονται περίπου σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ 4 δηλαδή τις 100 των συνολικών συνεισφορών το τρίτο νέο στοιχείο είναι οι λεπτομερείς πληροφορίες και συγκρίσεις μεταξύ χωρών μελών που παρέχονται τώρα όσον αφορά τις ληφθήσεις πληρωμές και τις εφαρμοστήσεις δημοσιονομικές διορθώσεις. Με αναγνώριση και της περιπλοκότητας του προϋπολογισμού αλλά και των νέων στοιχείων που έχουν εισαχθεί, η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί και να συζητήσει περαιτέρω με την, Κομισιόν, με την Επιτροπή σας και να δώσει και άλλες εξηγήσει. Ευχαρίστως λοιπόν να οργανώσουμε ένα εργαστήριο για το θέμα. Εν τέλει, επιθυμώ να τονίσω ότι η Κομισιόν μπορεί να καταδείξει ότι έχει αποτελεσματικά δράση με μέτρα για να προστατεύσει τον προϋπολογισμό από παράνομη χρήση. Γνωρίζει την ε, πολιτική ευαισθησία του εγγράφου η Κομισιόν που θα υποβάλλεται κάθε χρόνο από εδώ και μπρος. Πιστεύει ότι η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντική συμβολή και για το 2012 αλλά και για τις συζητήσεις των μελλοντικών απαλλαγών. Τώρα ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που θέσατε κύριε Πίπερ για την Ισπανία και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έγιναν στην περίπτωση της χώρας αυτής. Το σημαντικό ποσό των διορθώσεων αυτών έχει σχέση με το, με το κλείσιμο της περίοδου, προγραμματικής περίοδου του 2006. Και οφείλει να λάβει κανείς υπόψη ότι υπάρχει μέσα στην διαδικασία μια λυσίδα ελέγχων και στην τελική φάση οι υπηρεσίες μας ελέγχουν με μεγάλη λεπτομέρεια όλες τις πληρωμές που έγιναν προς τους δικαιούχους, προς τις χώρες μέλη και εάν διαπιστώσουν οποιασδήποτε παρατυπίες στις δαπάνες επιβάλλουν δημοσιονομικές διορθώσεις στις χώρες αυτές. Στην δε περίπτωση της Ισπανίας διαπιστώθηκαν σημαντικές ανεπάρκειες του συστήματος για την περίοδο 2000-2006, κάτι το οποίο οδήγησε σε υψηλό επίπεδο δημοσιονομικών διορθώσεων για την περίπτωση της Ισπανίας. Σημαντικό ωστόσο είναι πώς ερμηνεύουμε τα ποσά αυτά. Ο στόχος μας με την ανακοίνωση ήταν να καταδείξουμε ότι η Κομισιόν έχει διάφορα εργαλεία στη διάθεσή της και προληπτικού και διορθωτικού χαρακτήρα εάν διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά σε κάποια χώρα μέλος. Και στο προληπτικό σκέλος περιλαμβάνονται και οι διακοπές και αναστολές πληρωμών που είδατε ότι αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσά τους στην διάρκεια του 2012 αλλά το πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το πολυετές σύστημα ελέγχων είναι η έλεγχη εκ των υστέρων και οι δράσεις που αναλαμβάνονται εάν αυτοί οι εκ των υστέρων έλεγχοι εντοπίσουν προβλήματα στη χώρα μέλος. Με την υποβολή των αριθμητικών αυτών στοιχείων δείχνουμε ότι αν εξετάσει κανείς σε πολυετή βάση την εφαρμογή των προγραμμάτων μας, όπως έγινε και από τον δικό μας ελεγκτή, διαπιστώνουμε ότι προστατεύεται επαρκώς ο κοινοτικός προϋπολογισμός από εσφαλμένες δαπάνες, λόγω και του διορθωτικού σκέλους των ελέγχων μας. Και εντατικοποιήσαμε σημαντικά την χρήση του διορθωτικού σκέλους. Και όταν βέβαια επεμβαίνει το διορθωτικό σκέλος, τότε ζητείται από τη χώρα μέλος να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στο σύστημα ελέγχων της, στα συστήματά της, έτσι ώστε να αποφύγει τέτοιες εξελίξεις στο μέλλον. Και βέβαια υπάρχουν θέματα στην Ισπανία που έχουν σχέση και με τον υψηλό βαθμό αυτονομίας ε, που διαθέτουν ορισμένες περιφέρειες και στις δυσκολίες εφαρμογής διαφόρων κανόνων. Αλλά αυτό είναι βέβαια πολιτικού χαρακτήρα θέμα και έτσι είναι, δομημένη η, έτσι είναι δομημένο το βασίλειο της Ισπανίας και γίνονται και διαφορετικές ερμηνείες, δίνονται διαφορετικές ερμηνείες στις διάφορες περιφέρειες της Ισπανίας. Τώρα για την επιχρήσωση νομίζω ότι το κάλυψα το θέμα αυτό ε, στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Ένας ε, σημαντικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και μάλιστα δουλέψαμε πολύ σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. είναι να εισαγάγουμε απλοποιημένες μεθόδους υπολογισμού κόστους για, την δαπάνη, για τις δαπάνες ορισμένων προγραμμάτων, γιατί αυτό επιτρέπει να αποφύγουμε την περιπλοκότητα των κανόνων και να μπορούμε να δίνουμε κατά ποσά για συγκεκριμένα προγράμματα χωρίς πολύ βαριά κριτήρια επιλεξιμότητας και δεσμευτήκαμε κιόλας να υποβάλουμε εκθέσεις για την κατάσταση της επιχρήσωσης gold plating στις διάφορες χώρες μέλη, ώστε να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες περιπτώσεις σε ορισμένες χώρες μέλη. Και αυτή νομίζω είναι η σημαντική εξέλιξη την οποία προβλέπουμε σε σχέση με την νέα προγραμματική περίοδο όπου θα ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να υποβάλουν στην Κομισιόν σχέδια κανόνων επιλεξιμότητας για να δούμε αν οι κανόνες αυτοί ενδεχομένως προκαλούν ε, περιτά κολλήματα εντός των χωρών μελών λόγω ε, από πυρών ε, επιχρήσωσης. Αναφερθήκατε και σε άλλα κράτη-μέλη, στην Ελλάδα, την Ιταλία και άλλους. Νομίζω ότι ένα υψηλό επίπεδο διορθώσεων που έχουν γίνει απέδειξε ότι εμείς μπορούμε να δράσουμε στα κράτη-μέλη όταν εντοπίζουμε προβλήματα με τα κοινωνικά κονδύλια και τελικά προστατεύουμε με αυτές τις δημοσιονομικές διορθώσεις ε, τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Γιατί οι διορθώσεις αυτές ε, εξαιρούνται των δηλώσεων πληρωμών και των αντισταθμίσεων και των ποσών τα οποία ε, θα γίνουν τελικά αντικείμενο ε, τέτοιου είδους διορθώσεων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο λοιπόν αυτές οι διορθώσεις που θα μας επιτρέψουν να προστατεύσουμε καλύτερα τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά με ex post ελέγχους στα πλαίσια του πολιετούς συστήματος ελέγχων γενικά. Ευχαριστώ Επίτροπε Σέματα. Ε, Έχω καιρό να δω μια τέτοια συζήτηση με τέτοιο ενδιαφέρον και τόσο σημαντικές εξηγήσεις από πλευράς της Επιτροπής και του Επιτρόπου. Let me say that we have a third group of Έχουμε μια ομάδα επισκεπτών που παρατηρούν Τις ε, εργασίας μας, τους καλωσορίζουμε και τώρα θα δώσω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο. Η εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον κύριο Σέμετα για τις συνοπτικές του εξηγήσεις. Μετά από τη διαδικασία απαλλαγής του 2011 βρήκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει ένα έγγραφο θα έλεγα αρκετά χρήσιμο. Ε, δεν μπορεί να συμφωνεί μάλλον με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου εκτός από τα σημεία όπου υπάρχει νομική αν θέλετε δυσκολία για να γίνουν δεκτές αυτές οι απόψεις. Εκπληρούν λοιπόν τις ε, απόψεις και τις προϋποθέσεις του Κοινοβουλίου το οποίο είναι υπεύθυνο και νομικά εφόσον υπάρχουν περιορισμοί νομικοί για τις συμφωνίες αυτές. Επίσης το θέμα των λαθών στις δημόσιες προμήθειες είναι ένα βασικό πρόβλημα σε σχέση με τις κοινοτικές δαπάνες, όπου παρουσιάζονται λάθη. Το θέμα των επιδόσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια ε, της ε, ε, οικονομικής διαχείρισης. Ε, η επόμενη περίοδος δαπανών 14 με 20 παραμένει ε, κυρίως συγκεντρωμένη στο θέμα των εσόδων και αυτό είναι μια ειδική δυσκολία και για τον έλεγχο των υστέρων αλλά και ε, για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σχολιάσω επίσης και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Οι επιστροφές ε, πραγματικά καλύπτουν πάρα πολύ υψηλά ποσά. Οι ανακτήσεις ποσών ε, για το 12 ήταν σε ε, ύψος ε, ιδιαίτερα μεγάλο όπως αν προσθέταμε τις αντίστοιχες επιστροφές από το 2006 και για αρκετά χρόνια. Υπήρξαν πάρα πολύ, πολλά λάθη ιδιαίτερα στον τομέα των πληρωμών συνοχής. Υπάρχουν αρκετές πλευρές τις οποίες μπορούμε να ελέγξουμε για περισσότερα λάθη στον τομέα των δαπανών. Ε, οι δαπάνες αντικατάστασης επηρεάζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς περισσότερο παρά υποχρεωτικά τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό το οποίο δεν φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι οι αναπληρωτικές αυτές δαπάνες δεν οδηγούν σε νέες μορφές δαπάνης χωρίς λάθη οι δαπάνες αντικατάστασης οι οποίες γίνονται πολλές φορές προγραμματικά σε σύντομους χρόνους στο τέλος της περίοδου εκτέλεσης του προγράμματος παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους και σε επίπεδο διαχείρισης και σε επίπεδο ελέγχων. Δεύτερη παρατήρηση στα πλαίσια αυτής της κριτικής ανάλυσης την οποία κάνω αναφέρεται στις οικονομικές αυτές διορθώσεις. Πολλές φορές δεν φτάνουν σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης των δαπανών και δεν καλύπτουν όλα τα λάθη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει βέβαια για αυτές τις διορθώσεις, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη ε, να ε, είναι υπεύθυνα για την ανάκτηση. Μερικές φορές γίνεται αυτό και αυτό οδηγεί συχνά σε πολύ ε, χαμηλά ποσοστά λαθών. Αυτό δεν γίνεται βέβαια πάντα γιατί τα κράτη-μέλη αποφασίζουν διαφορετικά. Εάν ένα κράτος ε, μέλος δεν ε, αποδίδει, αυτό σημαίνει ότι ο ένας από τους διαχειριστές δεν αποδίδει και τα λάθη παραμένουν τελικά σε σχέση με τις πληρωμές στη συνοχή. Ε, να μην ξεχνάμε ότι για τις οικονομικές αυτές διορθώσεις και τις ανακτήσεις απαιτείται συνεργασία όλων των πλευρών. Η έκθεση εν πάση περιπτώσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ε, δρά γρήγορα πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλύτερα ενήμερη για το ποια είναι η κατάσταση που ισχύει, αλλά αυτό δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα σε επίπεδο προγραμμάτων. Ε, το συνέδριο ήδη από το 2009 στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσή του τα είχε ε, υπογραμμίσει όλα αυτά και για το 12 οι αναλύσεις αυτές θα επαναληφθούν. Βασίζονται σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή χρησιμοποιεί και αυτή τα ίδια δεδομένα σχετικά με τις ανακτήσεις και διορθώσεις. Ακόμα λοιπόν και η έκθεση αυτή έλθει δημοσιευθεί μετά τη δημοσίευση της έκθεσής μας για το 12 η θέση μας περιλαμβάνεται έτσι και αλλιώς στο κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσης του συνεδρίου ή ε, επίσης εκθέσεις ετήσιας δραστηριότητες, όπως επίσης και οι δραστηριότητες των εσωτερικών ελέγχων για την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλυφθεί ε, στην ε, ετήσια έκθεση του συνεδρίου για το 12 και αυτό με περιορίζει να μιλήσω περισσότερο σήμερα. Τώρα σε κάποιες συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις που τέθηκαν ε, από τον εισηγητή που είναι ε, και για μας θέμα. Πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία ανάκτησης πιο ουσιαστική και αποτελεσματική. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περισσότερα κίνητρα για τη διαδικασία αυτή και εφόσον τα ποσά τα οποία δηλούνται ε, χαρακτηρίζονται από λάθη και φύγουν τα λειτουργικά προγράμματα θα πρέπει να ελέγχονται από τα ίδια τα κράτη καταρχάς. Θυμίζω ότι επανειλημμένα στην έκθεση μάλιστα για το 12 το ελεγκτικό συνέδριο έχει διαπιστώσει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ανοιχνεύσουν και να διορθώσουν τα λάθη επί τη βάση των αρχικών εγγράφων που προώθησαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είχαν κάνει τους ελέγχους αυτούς. Αυτό επαναλαμβάνεται δυστυχώς σε αιτήσια βάση και φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη βούλησης εντοπισμού και διόρθωσης των λαθών πριν παραπέμψουν τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να αλλάξει για να γίνει η διαδικασία ανάκτησης και διόρθωσης ταχύτερη. Ευχαριστώ. Τρεις ομιλητές έχω που ζητούν το λόγο, ο Ντέρκ Βον, η κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Γκάιερ. Με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο, αυτή είναι η σειρά, ο κύριος Ντέρεκ Βον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσίασή του, αλλά και το Ελεκτικό Συνέδριο, καθώς επίσης και τον εισηγητή για τις τοποθετήσεις του. Ε, Χαίρομαι για, και καλωσορίζω για τη συνθετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ανακοίνωση για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά. Όταν γίνεται πρόοδος και δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι έχει γίνει, καλό είναι να το αναγνωρίζουμε ε, όταν το παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λέω με σαφήνεια. Κάτι άλλο που επίσης θεωρώ σημαντικό θέμα είναι το εξής. Εμείς θέλουμε να ε, ονόμαστε ε, ότι ε, γίνεται σωστή δαπάνη των πόρων και κατά την άποψή μου η λιτότητα ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα. Γιατί πραγματικά κάθε ευρώ που χρησιμοποιείται σωστά, που πιάνει τόπο, βοηθάει να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Οπότε κάθε ευρώ μετράει ή θα έπρεπε να μετράει. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν τη θετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για κάποιες μεθόδους απλούστευσης που προτείνει ε, για την επόμενη περίοδο μέχρι το 2020 και στη συνοχή και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα απλουστευτικά μέτρα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους νομοθέτες και υπενήσεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Μα δεν νομίζω. Ε, το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την ηλεκτρονική συνοχή, το e και τους κοινούς κανόνες των πέντε ταμείων ε, των βασικών της συνοχής. Για κάτι που αναφέρατε κι εσείς, κατά αποκοπή, ποσά ή πληρωμές. Και εμείς είμαστε υπέρ της απλούστευσης στο μέλλον. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει και τα κράτη-μέλη να ε, το λάβουν αυτό το μήνυμα για να είναι ε, πιο απλές οι διαδικασίες για εκείνους που υποβάλλουν αίτηση. Γιατί τα σφάλματα που εντοπίζονται από το ελεκτικό συνέδριο και στο παρελθόν και τώρα και από εσά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία από τις πηγές ε, προβλημάτων ήταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η αδυναμία τήρησης τους ε, κατά την υποβολή της αίτησης ε, για τη χρηματοδότηση, για τους διαγωνισμούς, ας πούμε στους σπόρους του κοινωνικού ταμείου. Και στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αυτά και να γίνεται πλούστευση ε, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Χαίρομαι και για τα όσα εξαγγέλλεται για τις επιδόσεις και τις αποδόσεις των κρατών μελών και το ρόλο του, Το είπε και ο εισηγητής στην αρχή. Ε, παράδειγμα, στην έκθεσή σας αναφέρεται η εστίαση που πρέπει να δοθεί σε κάποια κράτη-μέλη στη Γεωργία που είναι πάνω από 2% το σφάλμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα ταμεία της ε, συνοχής. Μιλούμε για διακοπές, για αναστολές πληρωμών και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κοινωνικό ταμείο και το περιφερειακό ταμείο, αλλά δεν έχουμε λεπτομέρειες. Τι σημαίνει αυτό. Ε, ποτέ δεν έχουμε τα στοιχεία και είναι δύσκολο να φτάσει κανείς σε πληροφορίες. Θα μπορούσαμε στο μέλλον ίσως να έχουμε πιο διαφανείς διαδικασίες και μεγαλύτερη πληροφόρηση για την αεροστολή πληρωμών ή τη διακοπή ε, προγραμμάτων, ιδιαίτερα στα διορθωτικά ταμεία. Ως προς την απαλλαγή και τη σχετική έκθεση για φέτος, καλό θα ήταν και θέλω να συνεχίσω τη δουλειά που έχει αρχίσει ο συνάδελφος Γιάννης θα πρέπει να δούμε πού γίνονται τα σφάλματα, να ξέρουμε και τα σωστά διδάγματα και συμπεράσματα για το μέλλον, για να έχουμε βελτιώσεις και να προλαμβάνονται αυτά τα σφάλματα. Οπότε και σε αυτή την έκθεση της απαλλαγής, ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και Κοινοβούλιο κάνουμε κάποιες προτάσεις. Παράδειγμα, υποστήριξη ε, των αρχών, των διαχειριστικών και των ελεκτικών των κρατών μελών για να εντοπίζουν συστημικά ασφάλματα, να δίνουμε κάποιες οδηγίες, μια καθοδήγηση στις αρχές αυτές για ε, την απλούστευση. Εσείς θα μπορούσατε ως Επίτροπος να σχολιάσετε αυτές τις βελτιώσεις που έχουμε προτείνει και στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ασχοληθώ και με τα τρία έγγραφα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και μάλιστα σε κάποιο βάθος. Το ένα αφορά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανακτήσεις. Θα πείτε και άλλα, ε, είναι πολύ νωρίς, όχι, όλα μαζί, ωραία. Αυτό το έγγραφο με το παράρτημά του πραγματικά υπολείπεται το προσδοκιό μου πρέπει να σας πω και κατά πολύ. Μας λέτε για πρώτη φορά ποια είναι τα νέα στοιχεία. Ευχαριστώ που μας τα παρουσιάζετε. 3,2% ανάκτηση. Σιγά τα λεφτά. Είναι πολύ πιο ακριβό να έχεις ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για να εισπράττει ε, αυτές τις πενταροδεκάρες υπάρχουν ελλείμματα στο σύστημα και φταίει και η νομοθεσία βέβαια αλλά και η εφαρμογή. Ήδη από το 1994 τρία κράτη πρωτοστατούν, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Στη νέα περίοδο η Τσεχία ε, ξεπέρασε την Ιταλία, αλλά παραμένει η Ιταλία στα πρωτοκασάτα. Λοιπόν, αυτή η αδράνεια αυτή η εθελοτυφλία και η ε, κόλληση αργία με δυσαριστεί κύριε Επίτροπε. Κάθε χρόνο ε, ε, δίνει τις ευλογίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας λέτε πόσα είναι τα κράτη-μέλη και ποια και από πότε. Τώρα Βουλγαρία, Ρουμανία 2008, προηγουμένως επιφυλάξεις δεν μας την ανέφεραν καν και στα διαρθρωτικά ταμεία και στα γεωργικά. Τι να σας πω. Από ό,τι φαίνεται, κανένας από τους συναδέλφους σας δεν ρίχνει ε, ούτε ματιά αλλιώς. Θα πρέπει να πει κάποιος κάποια στιγμή, ας κάνουμε κάτι. Λοιπόν, μια που έλεγα ότι δεν το διαβάζει κανείς, να σας πω και κάτι άλλο. Μας φέρετε ένα έγγραφο για τις ανακτήσεις και πραγματικά με έχει κάπως πικράνει κάτι. Η σελίδα 21 και η σελίδα 36 ταυτίζονται. Άμα μας λέτε ε, όλα τα πράγματα δύο φορές, ωραία, έχουμε χοντρά βιβλία και τόμους, αλλά όχι ουσιαστικό περιεχόμενο. Για το έγγραφο εργασία έχετε βγάλει κάποια στοιχεία από εκεί για την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έχετε ξαναφτιάξει κάπω, αλλά το Staff Working Document είναι φωτοτυπία περίπου του εγγράφου. Και εγώ περίμενα λίγη περισσότερη προστιθέμενη αξία. Αν μου παίρνετε την νομοθεσία και την ξανατυπώνετε, τι να το κάνω. Να κάνω και μερικές ερωτήσεις τώρα. Πρώτον, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 τράβηξε λίγο τα λουριά, αλλά το ταμείο είναι μείον. Δεν έχουμε λεφτά οι πληρωμές δεν γίνονται. Πιέζουμε δηλαδή όταν στενεύουν τα πράγματα και δεν μπορούμε να κάνουμε τις πληρωμές μας. Αυτό είναι δραματικό, γιατί αυτό πραγματικά υπονομεύει και το νόημα των συστημάτων ελέγχου. Τι γίνεται στις χώρες της κρίσης από ανακτήσεις, τι επίκειται και τι εισπράτεται. Από τις τέσσερις χώρες που έχουν αναγκαστική διοίκηση που είναι σε προγράμματα, Στη σελίδα 27 αναφέρεται κάτι στο Staff Working ε, Document για τη δινή κατάσταση. Εντάξει, το ομολογείτε, αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να έχουμε μια εικόνα. Γίνεται λόγος για κάποια προειδοποίηση, για κάποια ε, ίσπραξη που αναμένεται, αλλά πότε. Καλό θα τα γνωρίζουμε αυτά. Και ποια είναι τα αποτελέσματα των ίδιων των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, έλεγχη των κρατών μελών, έλεγχη τη Επιτροπή. Πολύ ωραίος ο κατάλογος και σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά θα ήταν ε, χρήσιμο και σημαντικό να δούμε πώς λειτουργούν τα ελεγκτικά συστήματα, αν λειτουργούν στα κράτη-μέλη. Γιατί έχουμε πολύ διαφορετικά στοιχεία, από τα λίγα στοιχεία που έτσι κι αλλιώ διαθέτουμε, ε, να έχουμε άμεση σύγκριση θα ήταν χρήσιμο και σημαντικό να μας δώσετε κάτι τι έχει υπολογίσει ως φάλμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι έχουν υπολογίσει τα κράτη-μέλη με τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς για να μπορούμε και να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε αν λειτουργούν αυτά τα συστήματα τα ελεγκτικά στις χώρες. Έχω μια σειρά ερωτημάτων τώρα, ε, προκαταβολές, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσει αυτές τις παράλογες μεγάλες χρονικές περιόδους. Ενδιαφέρον το, το κείμενο, δεν λέω. 75% περίπου των προκαταβολών είναι πάνω από 18 μήνες ή πάνω από 6 χρόνια είναι 16 δις. Δηλαδή προκαταβάλουμε και μετά από 6 χρόνια τι να πούμε, πού είναι τα λεφτά, γιατί δεν έγιναν τα προγράμματα. Και τώρα δώσαμε και άλλη παράτωση. Μα τι καταστροφή είναι αυτή για την οικονομική διαχείριση. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η χρονική περίοδος και τι επιπτώσει έχει στην οικονομική διαχείριση αυτό. Θα πρέπει να ασχοληθεί καμιά φορά και ο εσωτερικός ελεγκτής με αυτό και να αποφανθεί. Γιατί είναι πραγματικός κίνδυνος όλη αυτή η περίοδος για τις ε, ε, πληρωμές που εκκρεμούν. Μόνο το 8% στα διαρθρωτικά ταμεία των προκαταβολών έχουν διεκπεριωθεί από το 2007. Πολύ προβληματικό αυτό. Έχω πολλές ερωτήσεις, τώρα δεν ξέρω τι να τις κάνω. Και για την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτού. Δραματική η έκθεση πεπραγμένων. Για τον εκτελεστικό οργανισμό ε, πολιτισμού, καλό θα ήταν να μας ενημερώσει. Έχουμε πολλές περιπτώσεις Όλαφ, 11 τον αριθμό και μία μιλάει για αυστηρές παρατυπίες ε, που έχει διαβιβαστεί στην Όλαφ το θέμα. Από πού έρχονται αυτά. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης διατείνεται συνεχώς ότι έχουν διαδικασίες και κατασκευές που ε, αποτελούν κίνδυνο ε, για τα οικονομικά. Θέλω να με ενημερώσετε και γι' αυτό, γιατί ακούμε διάφορα πράγματα ε, επίσης και από την Βουδαπέστη, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τεχνολογίας και θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ το πόρισμα του εσωτερικού οικονομικού ελέγχου. Θα τις ε, στείλω και γραπτός όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά υπάρχει ένα θέμα αρχής και ένα ερώτημα αρχής. Για ποιο λόγο παραμένουμε θεατές μέχρι να αντιδράσουμε και αντιδρούμε μόνο όταν μας τελειώνουν τα λεφτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης ε, Γκάιερ, παρακαλώ. Δεν έχω ερωτήσεις και μάλιστα τόσο πολλές και λεπτομερείς όπως η και Γκρέσλε. Με ενδιαφέρει πρώτα η κατάταξη αυτού του νέου εγγράφου. Ναι, μεν μπορεί να ασκήσει κανείς ε, για κάποιες λεπτομέρειες κριτική, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πρωτίστως είναι να τονίσω ένα θέμα. Επανέρχομαι και πάλι στον κύριο Μπονίτσι, πρώην μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, όπου ήμουν τότε νέος, νέο μέλος εδώ και σήκωσε ένα χαρτί και μας είπε τότε ότι μπορεί κανείς να διορθώσει σφάλματα με δύο τρόπους. Πρώτον, να βελτιώσει τα συστήματα ελέγχων, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, είπε, και ενθαρρύνουμε την Κομισιόν κάθε φορά που διαπιστώνει ότι τα συστήματα ελέγχου ε, λειτουργούν ανεπαρκώς να διακόψει ή να αναστείλει τις πληρωμές. Τα νούμερα αυτά αυξάνουν. Οφείλουμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι η Κομισιόν αντιδρά, όπως το ζητήσαμε. Η άλλη δυνατότητα που είχε τότε εξηγήσει ο κ. Μπονίτσι είναι να διορθώσουμε τα σφάλματα φροντίζοντας ώστε οι εσφαλμένες πληρωμές να μεταφέρονται σε νόμιμα προγράμματα ή να αφαιρούνται. Εγώ όταν εξέτασα το έγγραφο αυτό, η ιδέα που είχα ήταν να κάνω μια σύγκριση. Τα ποσοστά σφαλμάτων που εμείς, τέλος πάντων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εγώ δεν ήμουν ακόμη μέλος, βρήκαμε στην τελευταία ε, περίοδο πώς έχουν εξελιχθεί όσον αφορά τις διορθώσεις και τις ανακτήσεις. Ήταν μια ιδέα αυτή. Και καταλήγω να πω ότι ναι, εφόσον ε, δούμε, ο κύριος Πίπερ σωστά τόνισε πόσο μεγάλα είναι τα νούμερα αυτά, ότι λειτουργούν, αποδίδουν αυτές οι ανακτήσεις σε αυτά τα ύψη, αυτό σημαίνει τότε ότι είναι, έχουν γίνει διορθώσεις παράτυπων πληρωμών σε αυτή την έκταση. Άρα αυτό εμένα με ικανοποιεί ότι δηλαδή η Κομισιόν στον ρόλο αυτών που της αρμόζει του θεματοφύλακα των συνθήκων κάνει τη δουλειά της. Ναι, είναι ίσως έχεις δίκιο, όχι ακόμα όσο πρέπει και τι άλλο θα έπρεπε να γίνει και αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά αυτό που πρωτίστως διαπιστώνω εδώ είναι ότι σφάλματα που πολλοί από εμά έχουμε ε, διαπιστώσει μετά από ανάλυση των ετησίων εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου και που διαπιστώνουμε υψηλό αριθμό σφαλμάτων, βέβαια μπορεί να το δει κανένα τον αριθμό αυτού και μέσα στην ιστορική εξέλιξη, ότι διορθώνονται. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, το ελεγκτικό συνέδριο με το οποίο είχα την ευκαιρία να συζητήσω λέει ναι μεν αλλά δεν μπορεί, δεν είναι και τόσο εύκολο να συμψηφιστεί με τον υψηλό αριθμό των σφαλμάτων, διότι δεν συμπίπτουν ακριβώς οι ανακτήσεις με τα σφάλματα. Σωστό και ε, το κατανοώ. Σωστό, μεν, αλλά και συνηθισμένο επιχείρημα λογιστών ελεγκτών. Και Πώς να πάω εγώ τώρα στους φορολογούμενους ψηφοφόρους μου και να τους πω ότι προστατεύεται επαρκώς ο προϋπολογισμός της Ένωσης ή πάντως η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί. Δεν έχω φτάσει να πω ότι ναι, όντω έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι τα φοβόμασταν και αυτό είναι μια καλή είδηση. Νομίζω ότι η κατάσταση στην Ισπανία χρειάζεται ίσως προσεκτικότερη εξέταση. Έχουμε θίξει την κατάσταση αυτή στην Επιτροπή μας και άλλες φορές και σε δήλωσή του ο κύριος Σέμετα έχει πει ότι το πρόβλημα αυτό συνάπτεται και με την περιφερειακή δομή του Ισπανικού κράτους όπου φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες για το ποιος είναι υπεύθυνος για ποια πράγματα σε αυτή την περιφερειακή δομή ποιος ε, συντάσσει τα διάφορα σχέδια, ποιος φροντίζει και επιτηρεί την εκτέλεσή τους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Ισπανικές αρχές επιτρέπουν να εξαφανίζονται τα λεφτά με τέτοιο ανέμελο τρόπο. Πρόκειται για σφάλματα. Τα σφάλματα όμως είναι εκπληκτικά υψηλά. Θα δούμε τώρα και με τους συντονιστές. Θα συζητήσουμε και για τις αντιπροσωπείες και πού θα ε, τις αποστείλουμε και μέχρι τις εκλογές. Αλλά και για μετά τις εκλογές πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό ε, της Ισπανίας και πώς, ότι πρέπει δηλαδή είναι σίγουρο να μειωθούν τα σφάλματα. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Λιμπεράτσκι. Επιτρέψτε μου κύριε ε, Επίτροπε να σας παρακαλέσω να σχολιάσετε τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων μου. Άκουσα ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τους γενικούς ελέγχους και τους ειδικού ελέγχους οι οποίοι έγιναν από τον εσωτερικό μας ελεγκτή ο οποίος είναι μαζί μας εδώ και δεν ξέρω αν θα ήθελε ο ίδιος να αναφερθεί στα συγκεκριμένα θέματα, στους συγκεκριμένους ελέγχους που έγιναν για το ΦΠΑ και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, στις πληρωμές. Και μετά θα συνεχίσω εγώ με κάπως πιο γενικά θέματα. Okay, yes, please. Ε, εντάξει, σας παρακαλώ, αλλά μη μακρηγορήσετε, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση της κυρίας Γκρέσπε. Κατάλαβα τη μία από τις δύο μάλλον. Που αφορά το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεχνολογίας της Βουδαπέστης. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν μία αποστολή ελέγχου, η οποία ολοκληρώθηκε τελικά τον μήνα Απρίλιο και έκανε ορισμένες συστάσεις, οι οποίες ε, είναι δημόσιες, διαθέσιμες. Περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της Βουδαπέστης, που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Οι συστάσεις αυτές έχουν γίνει αντικείμενο και ενός προγράμματος δράσης που έγινε δεκτό όχι μόνο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο αλλά και από το Συμβούλιο Διοίκησης. Και οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται και τις παρακολουθούμε από κοντά. Δεν μπορώ να σας δώσω στην παρούσα φάση άλλες λεπτομέρειες. Πάντως στα πλαίσια της απαλλαγής η Επιτροπή σας έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει το περιεχόμενο της έκθεσης επί τη βάση των ισχυουσών προβλέψεων για την επίδοση εγγράφων εμπιστευτικών γύρω από ελέγχους που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αλλά η άλλη υπηρεσία που είπατε δεν την κατάλαβα, πάνω στην οποία έχετε πληροφορίες για εσωτερικό έλεγχο. Αλλά μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ε, ερωτήσεις της κυρίας Γκρέσλε τώρα ή και αργότερα αν δεν υπάρχει χρόνος. Ο Επίτροπος θα είμαι σύντομος. Ξεκινώντας, να σχολιάσω αυτά που είπε η εκπρόσωπος του συνεδρίου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων σε ορισμένα θέματα, is uh, that is to protect uh, EU uh, Τα μέτρα λοιπόν τα οποία εμείς εφαρμόζουμε ή να, ζητάμε να εφαρμοστούν ε, αφορούν είτε σε διακοπή πληρωμών είτε σε ανακτήσεις ποσών και εκ των διορθώσεις. Είτε προβλέπουμε δηλαδή, προληπτικά παρεμβαίνουμε, είτε εκ των υστέρων διορθώνουμε. Αυτό λέγεται αναλυτικά στην έκθεσή μας. Οι κανόνες οι οποίοι ισχύουν επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να αντικαταστήσουν τα λανθασμένα προγράμματά τους με νέα προγράμματα αλλά το να υποθέσει κανείς ότι τα νέα αυτά προγράμματα εξ αρχής ε, θα έχουν λάθη είναι μια προκατάληψη. Ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα μαθαίνουν από τα λάθη τα οποία έχουν κάνει και θα υποβάλουν προγράμματα τα οποία να είναι ε, ελεύθερα των προηγούμενων λαθών για την αναδρομικότητα δεν είναι κάτι το καλό, αλλά είναι κάτι που επιτρέπεται όμως επί τη βάση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Και είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο πνεύμα των νομικών ρυθμίσεων και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να το κάνουν και το κάνουν. Ο νόμος αυτός έγινε δεκτός από τους συνομοθέτες, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο προτείνουμε με ξεκάθαρο τρόπο η αναδρομικότητα να εξαφανιστεί από το σύστημα και ελπίζω η πρόταση αυτή να γίνει δεκτή. Όταν υπάρξει η τελική συμφωνία για τα θέματα των κανονισμών της πολιτικής συνοχής, όταν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία. Αντίστοιχο θέμα είναι αυτό που συνδέεται με τις ε, τελικές διορθώσεις, καθαρές διορθώσεις ε, υπό τους παρόντες ε, θα έλεγα ισχύοντες κανόνες δεν μπορεί να γίνουν τέτοιου είδους διορθώσεις. Αν στο τέλος της περίοδου το συνολικό ποσό είναι υψηλότερο από τα προγράμματα των κρατών μελών, αυτό οδηγεί στην τελική εκ των υστέρων διόρθωση αλλά όχι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ε, της διάρκειας του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το θέμα της πρόληψης σε σχέση με την εκ των διόρθωση που τέθηκε και από την κυρία Γκρέσλα. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε βέβαιοι ότι ένα επαρκές επίπεδο πρόληψης εφαρμόζεται με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, με την διακοπή των πληρωμών προσωρινή μη και με τα υψηλά ποσά τα οποία βλέπουμε στην έκθεση, εμείς χρησιμοποιούμε τελικά αυτό το προληπτικό κομμάτι όσο μπορούμε περισσότερο. Εάν όμως ε, διαπιστώσουμε εκ των υστέρων κάποια λάθη, είναι καθήκον μας να τα διορθώσουμε τα λάθη αυτά. και ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών της Επιτροπής ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια γύρω από αυτό. Ενθυμίστε ότι στα πλαίσια του νέου κανονισμού του δημοσιονομικού θα πρέπει να παρουσιάσουμε επίσης και πρόβλεψη κόστους ελέγχου όταν κάνουμε νέου τύπου προτάσεις νομοθετικές. Είμαστε λοιπόν στην διάθεσή σας έτσι ώστε να σταθμίσουμε εν πάση περιπτώσει το σε τι ανταποκρίνεται το κόστος του ελέγχου στα αποτελέσματα δηλαδή που αναμένουμε από τους ελέγχους αυτούς. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με τη νέα ρύθμιση θα έχουμε μια πιο διαφανή κατάσταση σε σχέση με το κόστος των ελέγχων και τις επιπτώσεις του κόστους στην ε, ε, σωστή οικονομική διαχείριση. Το θέμα της έλλειψης χρημάτων και αν είναι λόγος για την ε, εντατικοποίηση της προσπάθειας την οποία κάνουμε. Όχι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες. Αυτό εφαρμόστηκε και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων απαλλαγών. Εμείς εντατικοποιούμε τις δραστηριότητές μας και σε προληπτικό επίπεδο και εκ των υστέρων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε πλήρως τις συστάσεις αυτές, κάτι το οποίο οδήγησε στην σημαντική αύξηση των διορθώσεων, των οικονομικών, των διακοπών πληρωμών προσωρινών ή τελικών. Σχετικά με τα μέτρα απλοποίησης τώρα, θέμα το οποίο τέθηκε από αρκετούς, γνωρίζετε ότι έχουμε προτείνει κύριε Βον ένα πακέτο προτάσεων απλοποίησης για το επόμενο FFM. Δυστυχώς πολλές από τις προτάσεις αυτές έχουν ε, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εξαφανιστεί στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και αυτό είναι κρίμα. Εδώ τίθεται το θέμα των συνομοθετών που θα πρέπει να βρούνε κάποιες προτάσεις, να καταλήξουν σε κάποιες προτάσεις κοινέ. Εμείς παρουσιάσαμε μια ειδική ανακοίνωση για τα θέματα της απλοποίησης. Προωθήσαμε την ιδέα της απλοποίησης όσο μπορούσαμε περισσότερο με συγκεκριμένα μέσα που θα οδηγήσουν σε μέτρα που ε, εφαρμόζουν απλοποιημένες διαδικασίες. Όπως είπε και η εκπρόσωπος του συνεδρίου, εάν οι διαδικασίες είναι απλούστερες, αυτό θα οδηγήσει και σε χαμηλότερα επίπεδα λαθών. Δυστυχώς, όταν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, οι καλές ιδέες δεν αρκούν. για το θέμα της μεγαλύτερης διαφάνειας, για τις διακοπές προσωρινές τελικές. Το σημείωμα υπαρίθμου 6 της ετήσιας έκθεσης παρουσιάζει έναν κατάλογο των κρατών μελών όπου έχουν σημειωθεί διακοπές προσωρινές και τελικές θα λοιπόν πληρέστατη σε επίπεδο διαφάνειας και αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και πληροφορίες θα το εξετάσουμε. Πάντως μπορούμε εμείς να σας παραπέμψουμε στα στοιχεία τα οποία ήδη έχουμε κυκλοφορήσει που αφορούν τους ετήσιους λογαριασμούς της τη λογιστική χρήση συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, μία ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε σχετικά με τις χώρες σε πρόγραμμα. Ε, ε, εννοήσατε ότι εμείς έχουμε χαλαρώσει τους, ε, την αυστηρότητά μας στις χώρες αυτές. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εφόσον υπάρχουν παραβιάσεις των κανόνων, οι παραβάσεις των κανόνων στις χώρες που ακολουθούν πρόγραμμα παρά την δύσκολη κατάσταση, εμείς εφαρμόζουμε πληρέστατα τους ισχύοντες νόμους και σε προληπτικό επίπεδο και σε διορθωτικό εκ των υστέρων επίπεδο. Σχετικά με το θέμα αυτό, έχουμε ε, σαν παράδειγμα σταματήσει τις πληρωμές σε σχέση με το κοινωνικό ταμείο, με το περιφερειακό ταμείο που τέθηκε και από τον κύριο Πίπερ και άλλους. Όταν το μέσο αυτό τέθηκε στη διάθεσή μας, το κοινωνικό ταμείο Ε, είχε τύχει της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου αντίθετα με τα περιφερειακά ταμεία. Αλλά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους παραλληλήσαμε ουσιακά, ευθυγραμμίσαμε συγγνώμη να το πω καλύτερα τις διαδικασίες και έτσι τώρα και τα δύο ταμεία μέσω του κανονισμού τους εφαρμόζουν τους κανόνες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάτι το οποίο οδηγεί στην αύξηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται και στα περιφερειακά ταμεία και όχι μόνο στο κοινωνικό ταμείο όπως βλέπετε από τους αριθμούς της έκθεσης. Κλείνοντας τώρα. Κυρία Γκρέσλε είπατε ότι περιμένατε περισσότερα από την έκθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πω και εγώ προτείνω να οργανώσουμε μια ομάδα ή μάλλον ένα εργαστήρι συζήτησης και να δούμε από κοντά όλο το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας και να συζητήσουμε επίσης και κάποιες περαιτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον κριθεί ότι χρειάζεται. Γιατί κάποια από τα θέματα είναι πάρα πολύ περίπλοκα και νομίζω ότι μια τέτοια συνάντηση θα δημιουργήσει ε, προϋποθέσεις καλύτερης κατανόησης της δράσης μας στα πλαίσια της προστασίας του κοινοτικού προϋπολογισμού. Κάτι το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε μέσω της ανακοίνωσής μας. Είναι η πρώτη ανακοίνωση του είδους αυτού την οποία κάνουμε και είμαστε απόλυτα στη διάθεσή σας για τρόπους και προτάσεις βελτίωσης της ανακοίνωσης αυτής στο μέλλον. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάιερ για τα σχόλιά του. Ο κύριος Γκάιερ μας είπε ότι τα μέσα τα οποία είναι στην διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρησιμοποιούνται και όλο και περισσότερο. Φυσικά δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο, αλλά κάτω από το παρόν σύστημα ισχύων, σύστημα ελέγχων, μπορώ να πω ότι ο, κοινωνικός, ο κοινοτικός προϋπολογισμός προστατεύεται καλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Σιγητά, κύριε Πίπερ, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να κλείσω και να αξιολογήσω λίγο τη συζήτηση. Θέλω να πω στον κύριο Ταβέν ε, από τον εσωτερικό έλεγχο ότι θα σας στείλουμε γραπτά κάποιες ερωτήσεις γιατί δεν προλάβαμε σήμερα να τις ε, απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Επίτροπε, προτείνεται εργαστήριο. Ως εισηγητής δεν θα σας κάνω τη χάρη να μπούμε τώρα και να χαθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ε, ενημέρωση έχουμε αρκετή. Δεκαετίες τώρα ξέρουμε ότι κάτι πάει στραβά. Στις ίδιες πάντα χώρες. Και πολύ συνειδητά στην αρχή ερώτησα ε, ποια συμπεράσματα τώρα θα εξάγουμε. Προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε ότι υπάρχουν αυτόνομες περιφέρειες στην Ισπανία, αλλά για συνέπειες και συμπεράσματα δεν άκουσα τίποτα. Και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, αν τα κοιτάξουμε για την Ισπανία, πάλι στην ίδια κατεύθυνση πάει. Και βέβαια κάνουν ε, κάποιες κινήσεις, προσέχουν, λειτουργεί το σύστημα των διορθώσεων. Αλλά τόσα χρόνια χάνεται τόσο χρήμα, τόσο σκόπος, τόση τεχνογνωσία, τόση ενέργεια και αυτό είναι εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και περιμένουμε το αμέσως προσεχές διάστημα μία αντίδραση. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να υπάρξει βοήθεια σε αυτές τις χώρες. Σίγουρα θα ζητηθούν ε, ειδικέ έκτακτες ε, εκθέσεις για τις χώρες αυτές και από το ελεγκτικό συνέδριο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ζητήσουμε να ε, ε, πάει άμεσα στη διαχείριση των προγραμμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πιάνει πια η δικαιολογία ότι δεν έχουμε ε, το προσωπικό. Ο κύριος Μπαρόζο κάνει πολλές προτάσεις για το πού θα υποχωρήσει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οπότε θα πρέπει να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας. Αυτό που μας προτείνεται ως ε, εξήγηση δεν μας αρκεί. Και θα ήθελα να πω τέλος ότι σας προσκαλέσαμε σε μια ακρόαση το Νοέμβριο. επίσης σας προσφέρουμε δυνατότητες για ακρόαση. Αυτά είναι τα δικά μας εργαστήρια, αλλά δεν έχουν ακόμα ε, δεσμευτεί η Επίτροπη ή απαντήσει ότι θα έρθουν. Και θα υπάρξει και γραπτή συνέχεια τη σημερινή συζήτηση Δεν μας είπατε ποια συμπεράσματα προτείνετε, τι συνέπειες θα υπάρξουν. Όλο διαπιστώσεις είστε και εξηγήσεις. Εντάξει, αυτά τα ακούσαμε. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίπερ. Κύριε Πίτροπε, κυρίες και κύριοι, να κάνω μερικά σχόλια. Ο κύριος Γκάιερ αναφέρθηκε σε μια ιστορική στιγμή που είναι οι εκλογές. Και θα έρθουν οι εκλογείς μας να μας ρωτήσουν και πού είναι η αποτελεσματικότητα και απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό. Δεύτερον, το είπε και ο εισηγητής. Ζητούμε όλο και περισσότερο ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε και υπόλογοι. Κάθε πέντε χρόνια λογοδοτούμε και ε, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να είναι υψηλό ε, το επίπεδο σφαλμάτων, αλλά ε, οι υπάλληλοι σας δουλεύουν καλά. Επίσης, ποιες είναι οι διαφορές σας με το ελεκτικό συνέδριο, κύριε Επίτροπε. Από τη μια σημαίνει ότι είστε ανεξάρτητα σώματα. Εντάξει, αλλά τα στοιχεία που μας δίνετε δεν μπορεί να είναι διαφορετικά ή τα διδάγματα που εξάγεται από διάφορες ε, καταστάσεις δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και κύριε Επίτροπε, τι κάνετε, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει το τέλος της θητείας. πώς θα ασκήσουμε εμείς ε, την εξουσία του κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχουμε πέραν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλο και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παίρνει το ρόλο μιας κυβέρνησης, ας πούμε, ε, την αντιστοιχεία σε μια χώρα και το κοινοβούλιο ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι αξιόλογες οι προσπάθειές σας κύριε Επιτροπέ και τις εκτιμούμε, αλλά καμιά φορά θα πρέπει να κοιτάτε και τη δημιουργικότητα που εμφανίζουν ε, τα διάφορα κράτη-μέλη για να περιπλέκουν τις διαδικασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί πολλές φορές το παρακάνουν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και το ελεκτικό συνέδριο και τον κύριο σε μετά προσωπικά. Ε, Αγαπητή Κέρστη από το ελεγκτικό συνέδριο. Και ας περάσουμε τώρα αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε, αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, δηλαδή λέω. Αντιπροσωπεία στη Βουλγαρία στα πλαίσια ε, του παροπλισμού ε, του Κοσλοντούι και ε, της κοινοτικής χρηματοδότησης. Η κυρία Γκρέσλε, επικεφαλής ε,